Je vous propose de commencer. Καλησπέρα σας αγαπητοί φίλοι. Προτείνω να ξεκινήσουμε την απογευματινή μας συνεδρίαση. Η πρόεδρός μας ε, συμμετέχει σε άλλη συνεδρίαση αυτή τη στιγμή και με παρακάλεσε να την αντικαταστήσω. Έχετε λάβει τις αποφάσεις των συντονιστών και αν δεν υποβληθούν παρατηρήσεις θα θεωρήσουμε ότι εγκρίνονται οι συστάσεις και οι αποφάσεις των συντονιστών. Έχετε διορία μέχρι το τέλος συνεδρίασης για να υποβάλλετε παρατηρήσεις ή αντιρρήσεις. Απογευματινή ημερή σε διάταξη. Πρώτο θέμα, η πρόταση κανονισμού που τροποποιεί το κανονισμό 810 του 2009 που θεσπίζει ένα κοινοτικό κώδικα θεωρήσεων. Πρόκειται να γνωμοδοτήσουμε στην αρμόδια επιτροπή που είναι η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών. Η μας είναι ο κύριος Ιστβάνου Λεγή, αλλά πουσιάζει και θα τον αντικαταστήσει η κυρία Δεμόντε. Ευχαριστώ. Σε ό,τι αφορά το τουρισμό και τις μεταφορές, είχαμε στο παρελθόν ήδη πρόοδο με το προηγούμενο πακέτο θεωρήσεων που πρότεινε και την αναδιατύπωση του κώδικα για τις θεωρήσεις και πριν από μία τριετία τον θεώρησε. Η τρέχουσα πρόταση απλουστεύει τις ε, παρούσες διαδικασίες για την έκδοση θεωρήσεων βραχές διάρκειας και υπάρχει ισορροπία μεταξύ της ασφάλειας ε, και της ε, πολιτικής θεωρήσεων. Επίσης, θέλουμε να διευκολύνουμε τις διαδικασίες χωρίς θεωρήσεων, ώστε νομιμοποιούνται τις σου, χωρίς όμως ε, να περιορίσουμε την ασφάλεια. Επίσης θα αυξηθεί η απασχόληση στον κλάδο του τουρισμού. Θα μπορέσει έτσι η Ευρώπη να συνεχίσει να είναι υπερθμόν ένα τουριστικός προορισμός. Η πρόταση απλούστευσης της διαδικασίας ε, εξυπηρετεί όσου θέλουν ε, να πραγματοποιήσουν βραχία παραμονή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μειώνει το κόστος και τη γραφειοκρατία. Τώρα, να σας πω ποια είναι τα βασικά επιτεύγματα. Μειώνεται καταρχήν η προθεσμία για την διεκπαιρέωση και λήψη απόφασης από 15 σε 10 μέρες. Ε, εξασφαλίσει τη δυνατότητα υποβολή αιτήσεων θεώρηση σε προξενία άλλων χωρών τη Ευρωπαϊκή Ένωση, εφόσον το κράτο μέλο που είναι αρμόδιο για τη διεκπαιρέωση τη αίτηση θεώρηση δεν έχει παρουσία ούτε εκπροσωπείται. Απλουστεύονται τα έντυπα αίτηση και υπάρχει δυνατότητα διαδικτυακών εφαρμογών. Επίσης ε, χορηγείται στα εξωτερικά σύνορα, ε, υποβάλλεται έτσι στα εξωτερικά σύνορα και προκειμένου να προωθεί ο βραχυπρόθεσμο τουρισμό, ένα κράτο μέρο μπορεί να αποφασίσει να επιτρέψει προσωρινά την υποβολή αιτήσεων θεώρηση, ειδικά σημεία διέλευση των χερσαίων ή θαλάσσιων σύνορων, το πολύ 7 μέρε. Σε σύγκριση με την πρόταση που ψηφίστηκε στην Ολομέλεια και ακόμη και με τον αρχικό κώδικα θεωρήσεων, υπάρχουν ορισμένα αποτελέσματα τα οποία δεν περιλαμβάνονται στη νέα πρόταση Επιτροπή. Για παράδειγμα, η υποχρεωτική έκδοση θεώρηση πολλαπλών εισόδων μεταβάλλεται σε ένα παρερμηνευμένο κλιμακωτό σύστημα. Η έννοια τη θεώρησης περιοδία και η ιδέα τη παροχή βοήθεια στου επαγγελματίε του πολιτισμού και του αθλητισμού απουσιάζουν επίση. Όλα αυτά δεν δείχνουν μια θετική προσέγγιση απέναντι στο έτος πολιτιστικής κληρονομιάς. Τέλος, η υποχρεωτική αύξηση των τιμών της θεώρησης δεν είναι ούτε δικαιολογημένη, ούτε αιτιολογείται δεόντως. Ε, σε ό,τι αφορά τη μελέτη επιπτώσεων, ε, ε, θα πρέπει οι θεωρήσεις έχουν τη μεγαλύτερη αύξηση και σε απόλυτους όρους και σε ό,τι αφορά τα έξοδα. Ο αριθμός των αφήξεων ε, στις χώρες Σέγγεν έχει αυξηθεί κατά 175% από το 2009 έως το 2016 στα 37,8 εκατομμύρια, ενώ ο συνολικός αριθμός αφήξεων αυξήθηκε μόνο κατά 38%. Επιπλέον, σε απόλυτους αριθμούς, Είχαμε περίπου 11 εκατομμύρια αφήξεις από το 2016 από την Κίνα, 6,5 εκατομμύρια από τη Ρωσία, 3,1 εκατομμύρια από αφρικανικές χώρες και 2,4 εκατομμύρια αφήξεις από την Τουρκία σε τουριστικά καταλήμματα στο χώρο Σέγγεν. Όλα αυτά επαναλαμβάνω για το 2016. Μάλιστα έχω καταθέσει και τροπολογίες για να ε, διευκολύνω την περαιτέρω εφαρμόγη. Καταρχήν, αύξηση τη δυνητική περίοδου ισχύω τη θεώρηση πολλαπλών εσόδων έω 10 έτη για νόμιου ταξιδιώτε που πληρούν τι προποθέσει σύμφωνα με τα αισθήματα θεωρήσεων άλλων τρίτων χωρών. Ε, προτείνω τη διατήρηση τη ισχύουσα διάταξη του κώδικα σχετικά με μακρύτερε περιόδου ε, ισχύω για τι θεωρήσει ε, σε, ε, σε αντίθεση με το σύστημα το προτινόμενο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που είναι κλιμακωτό και το οποίο δεν αναμένεται να συμβάλλει στην αύξηση τη έκδοση θεωρήσεων. Επίση, διευκολύνεται η παράταση παραμονή νόμων ταξιδιωτών εντό του χώρου Σέγγεν με παράλληλη τήρηση των ορίων του εθνικού δικαίου. Επιτρέπω στου ετούντε να υποβάλουν τη θεώρηση σε προξενείο άλλου κράτου μέλου όταν το προξενείο του αρμόδιου κράτου μέλου απέχει τουλάχιστον 500 χιλιόμετρα από την κατοικία του. ιδιαιτερε μεγάλε χώρε επιτρέπω με τις τροπολογίες μου τη χρήση ενός ποσοστού της αύξησης ε, του τέλους για τους ετούντες θεώρηση με σκοπό τη στήριξη της αποκοινού πρόθεσης της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τον Τουρισμό. Και μάλιστα έχουμε ήδη εξαιρετικά παραδείγματα σχετικά. Περιμένω τώρα τα σχόλια και τις προτάσεις σας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Θα ακούσουμε τώρα τους σκιώδεις εισηγητές. Ο Δήμ, εκ μέρους του ΕΛΚ φαντάζομαι, έτσι. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Και εγώ έχω την τιμή να αντικαταστήσω εδώ την Κλαδιο Μοντέρο, η οποία αγκυμονούσα λύπη με άδεια εγκυμοσύνης. Είναι ένα ευαίσθητο θέμα αυτό. Και το 2014 το έχουμε ε, συζητήσει με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το θέμα αυτό της πολιτικής θεωρήσεων τότε είχε απορρίψει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στο μεταξύ φαίνεται ότι ως Ευρωπαϊκή Ένωση είμαστε πιο αυστηροί όσον αφορά την διάθεση θεωρήσεων. Στον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού είμαστε κάτω από το μέσο όρο. Όσον αφορά τη διευκόλυνση δηλαδή θεωρήσεων Βέβαια υπάρχουν διάφοροι παράγοντες που παίζουν ρόλο. Από τη μια έχουμε τους τουρίστες, από την άλλη μεριά έχουμε τους επαγγελματίες, ε, και άλλου. Δυστυχώ όμως στην Ευρώπη έχουμε να κάνουμε και κατά πολύ με το θέμα της μετανάστευσης, της ε, νόμιμης ή της παράνομης. Η κυρία Μοντέρο λοιπόν βρίσκει πως η νέα πρόταση αξίζει τον κόπο. Όμως έχουμε κάποιες παρατηρήσεις. Πρώτον, η ηλεκτρονική θεώρηση, η ηλεκτρονική αίτηση για θεώρηση διακανονίζεται επαρκώς. Διότι στον Καναδά, τις Ηνωμένε Πολιτείε και την Ανατολική Ασία υπάρχει η δυνατότητα να ζητήσει κανείς ηλεκτρονικά τη θεώρηση, αλλά υπάρχει και μια συνέντευξη επίσης. Αυτό διακανονίζεται πιο καλά από ό,τι στη δικιά μας την περίπτωση. Οπότε δεν ξέρουν πως τελικά η δικιά μας η μέθοδος θα είναι πιο δύσκολη. Δεύτερον, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πάνε σε διάφορες χώρες ε, με πλοίο, είτε ο είτε άλλοι ναυτικοί κλπ. που πρέπει να ζητήσουν θεώρηση. Και δεν είναι ξεκάθαρο για τους ανθρώπους αυτούς τι θα κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρθρο 36, α, της πρότασης, όπου αναφέρεται αριθμός μηνών που πρέπει να ακολουθήσει για κοινοποίηση κάθε χώρα. Και ρωτάω, δεν θα μπορούσε να είναι πιο ευέλικτο αυτό το μέτρο και μήπως η πρόταση του 2014 για αυτό το συγκεκριμένο σημείο ήταν προτιμότερη. Έπειτα υπάρχει και κάτι άλλο όμορφο, τουλάχιστον έτσι εγώ νομίζω, ότι τα έσοδα από τις θεωρήσεις να πηγαίνουν στον τουρισμό. Αυτό προτείνεται εδώ. Βέβαια στην πράξη πώς θα υλοποιηθεί κάτι τέτοιο. Αυτές είναι οι παρατηρήσεις λοιπόν της συναδέρφου Κλάουντια Μοντέρο. Και εύχομαι στον εισηγητή μέσω της Κλάουντια κάθε επιτυχία στην υπόθεση αυτή. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ δε. Κύριος Λοντόστρη, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ και ευχαριστώ τον εισηγητή για την εκπόνηση της γνωμοδότησης. Παρόλο που δεν... Παρόλο που συμφωνούμε με την διευκόλυνση της χορήγησης θεώρησης ε, στους νόμους ταξιδιώτες, ε, ιδιαίτερα για οικογενειακούς, επιστημονικούς, τουριστικούς, επιχειρηματικούς λόγους. Θέλουμε ε, αυτοί οι άνθρωποι να έχουν τη δυνατότητα να επισκέφτονται πιο συχνά την Ευρώπη. Και σίγουρα είμαστε σημαντικός α, ε, τουριστικός προορισμός ε, και κάτι τέτοιο αποφέρει και οικονομικά πλονεκτήματα στην οικονομία μας. Γι' αυτό και καλό θα ήταν να διευκολύνουμε την χορήγηση θεωρήσεων. Αλλά μην ξεχνούμε ότι ταυτόχρονα η Ευρωπαϊκή Ένωση υπόκειται τεράστιε μεταναστευτικέ πιέσει και οι διευκολύνσει στο σύστημα θεωρήσεων μπορούν πολύ συχνά να μετατραπούν σε κενά και παραθυράκια που θα επιδέχονται χειραγώγηση ή εκμετάλλευση. Πολύ προσοχή λοιπόν σε ό,τι αφορά τη μείωση της προθεσμίας για τη διεκπαιρέωση και ε, λήψη απόφαση από 15 σε 10 μέρες. Η συντόμευση αυτής της προθεσμίας δεν δικαιολογείται και δεν ε, έχει πλεονεκτήματα, ενώ δημιουργεί τεράστιο κίνδυνο. Έχει περισσότερους κινδύνους παρά πλεονεκτήματα αυτή η σύντμηση της προθεσμίας από 15 σε 10 μέρες. Επίσης, ε, είπαμε ότι καλό θα ήταν να μιμηθούμε κάποιους ε, άλλους εταίρους, όπως τους Αμερικανούς, ό,τι φορά τη διαχείριση τέτοιων θεωρήσεων. Μάλιστα, σχετικά έχουμε καταθέσει τροπολογίες, την 5 και την 7. Οι Ηνωμένε Πολιτείε έχουν ε, ένα πολύ αποτελεσματικό σύστημα χορήγηση θεωρήσεων και λαμβάνει πολύ σωστά υπόψη τις διάφορες πτυχές της μεταναστευτικής πολιτικής. Καμία διευκόλυνση που στόχο έχει την αύξηση του τουρισμού δεν θα πρέπει να μετατραπεί σε απειλή ή αύξηση του κινδύνου και άσκηση πιέσεων στη χώρα, στο χώρο Σέγγεν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Σλοτόφσκι. Σράντα, παρακαλώ. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Και, ευχαρι... και υποστήριζα την πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής που διευκολύνει την χορήγηση της θεώρησης. Ταυτόχρονα υποστηρίζω το σχέδιο γνωμοδότησης του εισηγητού που ακολουθεί την ίδια γραμμή με, αυτή της, ε, με, με αυτό της πρότασης Επιτροπής. Καλό θα ήταν να είναι στο δυνατόν πιο ομοιόμορφα τα έγγραφα που τεκμηριώνουν το αίτημα και να βελτιστοποιηθεί η χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας και κατά την διαγραμμική υποβολή της αίτησης αλλά και κατά τη διάρκεια ολόκληρης διαδικασίας για την εξασφάλιση θεώρησης. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Γνωτού, ΕΛΦ. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ η μεταρρύθμιση που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή του κώδικα θεωρήσεων είναι μια καταπληκτική έκπληξη. Δεν περιμέναμε ότι θα υπάρχουν ε, στοιχεία που θα ακολουθούσαν αυτό που έστωσε η ομάδα μου, δηλαδή ενίσχυση των στοιχείων ασφάλειας ε, υποστηρίζω λοιπόν τα δύο στοιχεία της έκθεσης, την ομοίωμορφη διαχείριση του συστήματος ε, είτε μεμονωμένης είτε πολλαπλής θεώρησης ώστε να αποφεύγονται οι καταχρήσεις όπως ε, το, η αναζήτηση του πιο ευνοϊκού καθεστώτος χορήγησης αλλά ταυτόχρονα και το ζήτημα της θεώρησης μπορεί να αξιοποιηθεί ως μοχλός εναντί εκείνων των κρατών που δεν επιδεικνύουν ε, ε, καλή βούλη σε σχέση με τον εντοπισμό και ανάκτηση των ε, υπηκόων που έχουν παράτυπα και παράνομα μπει και, και παραμείνει στο ευρωπαϊκό, στην ευρωπαϊκή επικράτεια. Επίσης ε, θα προτιμούσαμε να υπήρχε και μία άρση διακοπή δηλαδή της, ε, του καθεστώτος θεώρηση εναντί των κρατών αυτών, αλλά αυτό δεν το προβλέπει η έκθεση. Η ε, αντιμετώπιση των μεταναστευτικών ροών πρέπει να είναι ένα κύριο μοχλό τη πολιτική των κρατών μελών. Ωστόσο, γιατί πάντα υπάρχει το ωστόσο, αυτή η θεώρηση, τι νόημα θα έχει, το σύστημα των θεωρήσεων δηλαδή, αν δεν εγγραφεί σε ένα ευρύτερο πεδίο πολιτικής της ε, μετανάστευσης ώστε να σταματήσουν να προβάλλονται τα επιχειρήματα εκείνων που θέλουν να υποστηρίξουν ε, την άκρατη μετανάστευση ή εκείνοι από τους Ευρωπαίους πολιτικούς που θεωρούν ότι μπορούν να αντικαταστήσουν τον Ευρωπαίο πολίτη από άλλους ε, για λόγους ε, δημογραφικούς. Η θεώρηση προς τα αφρικανικά κράτη, παραδείγματι, που αποφασίστηκε στη Βαλέτα, στην Ευρωπαϊκή Συνοδοκορυφής. Θα ήθελα επίσης να αναφέρω τα εξής δύο φαινόμενα το πρώτο που αφορά τους ετούντε άσυλο που επιστρέφουν στις χώρες ε, προέλευσης τους, όπου υποτίθεται πως κινδυνεύει η ζωή τους. Εάν συμβαίνει κάτι τέτοιο πρέπει να απελάβνονται ή να απαγορεύεται η επάνωδός τους. Δεύτερον, και για όσους παραμένουν παράνομα στην Ευρωπαϊκή, Ευρωπαϊκή Επικράτεια μετά την εκπνοή της ε, Ευρωπαϊκής θεωρήση της Σέγγεν, πριν από 10 χρόνια ακόμη η γερουσία τη Γαλλία είχε

της συνοριοφυλακής της Γαλλίας είχε δηλώσει πως στην Αλγερία ήταν προφανές το ότι υπήρχε απάτη σε σχέση με τη χορήγηση θεωρήσεων σε Αλγερινούς και έτσι ανοίγω παρένθεση έρχονται με θεώρηση διαβατηρίων πολύ Αλγερινοί στη Γαλλία χωρίς όμως να ξαναφεύγουν ποτέ και είναι η δεύτερη ομάδα εθνοτική ομάδα σε παράνομη κατάσταση, μάλιστα αυτοί οι οποίοι υποτίθεται πως τιμούν τη Γαλλία. Και κάτι ακόμη που πρέπει να γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή που, που σοβεί επιδημία χολέρα στην Αλγερία πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί σε σχέση με τη χολήξη θεωρήσεων Σέγγεν. Ευχαριστώ πολύ κύριε Αγνωτού. Αν δεν θέλει κανείς άλλο το λόγο. Παρακαλώ την κυρία Σέρντσεν εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να λάβει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Καλησπέρα σας. Δύο λόγια μόνο εισαγωγικά για να αναπτύξω την πρότασή μας, την πρόταση του 2018 γιατί όντως υπήρχε και μια πρόταση του 2014 η οποία δεν έφτασε ε, μέχρι το στάδιο της υιοθέτησης για διάφορους λόγους κυρίω γιατί δεν συμφώνησαν, δεν μπόρεσαν να συμφωνήσουν οι συνομοθέτε και έτσι αποφασίσαμε να αποσύρουμε την πρόταση. Ε, κατόπιν και ε, εν ώψη της νέας κατάστασης όπως αυτή αναδείχθηκε τα τελευταία χρόνια σε σχέση με τη μεταναστεύση και την ασφάλεια αποφασίσαμε να αναπτύξουμε μια πιο στοχευμένη και συγκεκριμένη νέα πρόταση θεωρώντας βέβαια ότι διατηρούμε πάντα κάποιες από τις πτυχές που διευκολύνουν ε, την θεώρηση από αυτές που περιείχε η πρόταση του 2014 για τις οποίες δεν είχε εξασφαλιστεί με τυπική συμφωνία αλλά άτυπα φαινόταν ότι γίνονται αποδεκτές ή θα μπορούσαν ε, να γίνουν αποδεκτές ε, συγκεκριμένες πρόνοιες. Θεωρούμε μάλιστα ότι αυτή η θα μπορουσαν να γινουν αποδεκτες συγκεκριμενε προνοιες πρόταση δεν έχει κίνδυνο να δημιουργήσει ένα σύστημα προϋποθέσεων θεώρησης που θα ε, αποτελεί τροχοπέδι στον τουρισμό ή γενικά τα ταξίδια. Για όποιο λόγο. Η αύξηση κατά 20 ευρώ στο τέλος θεώρησης είναι πολύ μετριοπαθής. Άλλωστε στην μελέτη αντικτύπου εξηγήσαμε πώς καταλήξαμε στο ποσό αυτό, στην αύξηση αυτή. Επίση, την ε, αξιολόγηση αντικτύπου, δεδομένου ότι προσπαθούσαμε να καταλάβουμε τι κοστίζει σε ένα καθώ κράτο μέλο η διαχείριση μια αιτήσεω θεώρηση, που αποδείχθηκε δύσκολο εγχείρημα και περίπλοκο. Τα 80 λοιπόν ευρώ αντιστοιχούν από ό,τι βλέπουμε σε τέλη που θα ίσιαν εάν απλώς είχαμε παρακολουθήσει τον πληθωρισμό σε ευρωπαϊκό επίπεδο όλα αυτά τα χρόνια, από το 2006. Όταν είχε επιβληθεί ως τέλος το ποσό των 60 ευρώ. Άρα η αύξηση δεν θεωρούμε ότι μπορεί να αποτρέψει κάποιον που θα θέλει να ταξιδέψει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επισημαίνω ότι στόχος των ε, τελών δεν είναι η παραγωγή εισοδήματο για τον Ευρωπαϊκό Προπολογισμό ή τα κράτη-μέλη, αλλά να υποστηρίξει τι δαπάνε ε, και τη διαδικασία που έχουν τα κράτη-μέλη για τη διαχείριση των θεωρήσεων και έτσι πιστεύουμε ότι ε, αντιστοιχεί στο νόγκο εργασία που προκύπτει από τις υποβληθήσει ανά έτος αιτήσεις θεώρηση. δεν επαναφέρουμε την πρόταση για την ε, πολλαπλή υποχρεωτική θεώρηση που είχαμε το 2014, αλλά έχουμε ένα σύστημα κλιμακωτό, το οποίο επίσης ε, καταλήγει να καθιστά υποχρεωτικό, ύστερα από μια σειρά βημάτων, ε, να χορηγεί το κράτος, ύστερα από 3-5 χρόνια, την πολλαπλή θεώρηση. Αυτό ήταν ένα από τα εμπόδια που είχαμε αντιμετωπίσει το 2014. Τα κράτη-μέλη θεώρησαν ότι για ορισμένε χώρε μπορούσε να είναι πιο γενναιόδορη Η Ευρώπη, όπω η παραδείγματη αντί τη Ρωσία, από την οποία είναι περιορισμένο ο μεταναστευτικό κίνδυνο, ενώ για άλλε χώρε, στι οποίε οι συνθήκε διαβίωση, ε, απασχόληση και λοιπέ μπορεί να αλλάξουν ριζικά ενδέχεται να ε, προκύπτει πρόβλημα ή κίνδυνος ε, μεγάλων μεταναστευτικών ροών. Έτσι λοιπόν έχουμε ένα σύστημα κλιμακωτό προτείνει με, το, με τη νέα πρόταση που επιτρέπει την προσαρμογή ανάλογα με τις συνθήκες ε, που επικρατούν στη χώρα προέλευσης των ετούντων. Κάτι ακόμη. Διατηρούμε το προσωρινό σύστημα στα εξωτερικά σύνορα για τη χορήγηση της θεώρησης δηλαδή στα εξωτερικά σύνορα αλλά με ενισχυμένη την ασφάλεια για λόγους προφανείς. Εφόσον επιλέξουν την δυνατότητα αυτή που τους προσφέρεται τα κράτη-μέλη για κάποιες σύντομες ε, περιόδους προκειμένου να ενισχύσουν ε, τον ε, τουρισμό σε συγκεκριμένε περιοχές πρέπει να πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις. Επίσης, εάν πρόκειται να εισαχθεί αυτό το προσωρινό σύστημα, όλες οι προϋποθέσεις, οι όροι και η περιγραφή του συστήματος πρέπει να έχει κοινοποιηθεί εκ των προτέρων. Πράγμα το οποίο επίση απαραίτητο. Τα κράτη-μέλη ταυτόχρονα ομιλούν για περαιτέρω ψηφιοποίηση. Είμαστε ε, σε επιφυλακή για το θέμα αυτό και μάλιστα αν παρακολουθήσατε και την ανακοίνωσή μας από πέρσι είχαμε αναφέρει σε σχέση με την πολιτική για τη θεώρηση ότι είναι απαραίτητο να εισαχθεί κάθε μορφή νέας τεχνολογίας ώστε να διευκολυνθεί η διαδικασία της υποβολής αίτησης και διαχείρισης της αίτηση για τη θεώρηση. Κατά τα άλλα όμως υπάρχουν περιοχές στον κόσμο που δεν εξασφαλίζουν ευχερή πρόσβαση στις νέες τεχνολογίες. Άρα το σύστημα δεν μπορεί να είναι αποκλειστικό, αποκλειστικά ψηφιακό. Ωστόσο, έχουμε μια σειρά από μελέτε στη διάθεσή μα και περιμένουμε νέε που θα μα εξηγήσουν, θα μα δώσουν λύσει για το πώ μπορούμε να απαλλαγούμε από την επιχάρτου αίτηση. Ένα επιπλέον εμπόδιο δηλαδή που πρέπει να αντιμετωπιστεί, πρέπει να εισαχθεί το σύστημα, να διασφαλιστεί, να εξασφαλιστούν τα στοιχεία ασφαλείας του νέου συστήματο, αλλά ξέρουμε ότι κάθε φορά που γίνεται επικαιροποίηση των όρων ασφαλεία, πάντα κάποιο ε, πιο πονηρό θα μπορέσει να βρει τον τρόπο να τα καταστρατηγήσει. Άρα και αυτό πρέπει να το παρακολουθούμε. Πάντως αν προχωρήσουμε στην αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών με την ε, ψηφιοποίηση θα έχουμε λύσει πολλά ζητήματα και ταυτόχρονα δεν θα είναι απαραίτητη η πρόσβαση, η προσέλευση στο προξενείο προκειμένου να επιτεθεί η θεώρηση πάνω στο διαβατήριο. με το αυτοκόλλητο, δηλαδή θα μπορούσε, αν καταργηθεί το αυτοκόλλητο θα μπορούσαμε να, να λύσουμε έτσι πολλά άλλα συναφή προβλήματα. Αυτά όμως για το μέλλον. Πρόταση για το θέμα αυτό δεν πρόκειται να καταθέσουμε αυτή τη στιγμή. Περιμένουμε πρώτα τα αποτελέσματα των μελετών και θα επανέλθουμε. Ενδεχομένως με κάποιες νέες προτάσεις ως και την ε, αλλαγή της νομικής βάσης. Πάντως επιτρέπουμε με την νέα αυτή πρόταση στα κράτη-μέλη τη χρήση των διαγραμμικών πλατφορμών για τις αιτήσει θεώρηση. και για την ε, δυνατότητα ε, αποστολής με ηλεκτρονική μορφή σκαναρισμένου αντιτύπου των εγγράφων, ώστε να μην χρειάζεται η προσέλευση στο προξενείο. Αυτά και σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Σόρενσεν. Επανέρχομαι στην κυρία Ντεμόντε. Η συγγήτρια έχετε σχόλια. Ευχαριστώ πολύ για τις προτάσεις. Νομίζω ότι τα όσα ακούσαμε προσανατολίζονται στη βελτίωση της κατάστασης όσον αφορά την τουριστική θεώρηση για το τουρισμό είναι 10%. Και βέβαια υπάρχει και όλο το περιβάλλον ε, δραστηριοποίησης που θα πρέπει να έχουμε υπόψη ε, στις προσπάθειές μας για απλούστευση, επιτάχυνση και βέβαια και δυνατότητες που προσφέρει η ψηφιοποίηση και η καινοτομία δεν πρέπει να παραγνωριστούν. Όλα αυτά τα καταγράφω και τα παραπέμπω στο συνάδελφό μας με τις προτάσεις των συναδέλφων για να ακολουθήσει τη διαδικασία στην επόμενη φάση. Merci, Madame Leonté. Donc... Euh, Ευχαριστούμε. 11 Σεπτεμβρίου είναι η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών. Στην Επιτροπή μας θα ψηφίσουμε στις 9 Οκτωβρίου. Γνωμοδότηση επί της ουσίας στη Λίμπε στις 5 Νοεμβρίου θα γίνει η ψηφοφορία. Δεν ξέρουμε ακόμα πότε θα ψηφιστεί το θέμα αυτό στην Ολομέλεια, ίσως στα τέλη της χρονιάς. Και περνάμε τώρα στο επόμενο θέμα που είναι τα μία αρχή ευρωπαϊκή εργασίας. Είναι γνωμοδότηση στην Επιτροπή Απασχόλησης. Ο Μικαήλ Τεζάν έχει το λόγο τώρα. Παρακαλώ. Πρόεδρε, ε, χαίρομαι που έχω την ευκαιρία να παρουσιάσω είναι έκθεσή μου για την Ευρωπαϊκή Αρχή Ελέγχου στην Επιτροπή μας. Έχουμε να κάνουμε με ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα της, ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή την εσωτερική αγορά ε, που στηρίζεται σε διάφορους πυλώνες, μεταξύ των οποίων ο ανταγωνισμός ε, που εξασφαλίζει οι θεμητές συνθήκες ανταγωνισμού για τις επιχειρήσεις, και βέβαια ανοίγει και μια αγορά 500 εκατομμυρίων καταναλωτών. Όταν παραβιάζει κανείς αρχές του ανταγωνισμού, οι επαπειλούμενες κυρώσεις ανέρχονται μέχρι το 10% του κύκλου εργασιών. Ε, Ένα δεύτερο πυλώνα είναι το δίκαιο, το κοινωνικό και το εργατικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο όμως δεν έχει ακόμη αναπτυχθεί ε, όπως θα έπρεπε και όπως περιμένουν οι πολίτες. Αγαπητοί συνάδελφοι, λοιπόν, με απασχολεί ιδιαίτερα το ερώτημα γιατί να μην υπάρχει κύρωση και δίωξη βάρος ε, επιχειρήσεων οι οποίες παραβιάζουν την κοινωνική νομοθεσία. Εάν το δίκαιο του ανταγωνισμού είναι μια δεμόκλειος σπάθη για τις επιχειρήσεις αυτές, γιατί να είναι ένα κουταλάκι του γλυκού το κοινοτικό δίκαιο για τα ε, δικαιώματα των εργαζομένων και τα κοινωνικά δικαιώματα. Νομίζω ότι πρέπει να υπάρξει μια ανταλλαγή μεταξύ Ευρωπαϊκής Αρχής και Εθνικών Κρατών, Εθνικών Αρχών. Αυτή η αρχή, η ΕΛΑ, Ευρωπαϊκή Αρχή για, για την απασχόληση, μπορεί να έχει αρμοδιότητες σε διάφορους τομείς και το χώρο των μεταφορών οπωσδήποτε, όπως θα θέλαμε εμείς, Τρία πράγματα είναι πάρα πολύ σημαντικά. Καταρχάς, η φυσταμένη κοινοτική νομοθεσία για το τομέα των μεταφορών με βάση την Οδηγία 561 του 2006, όπου προβλέπεται πως ε, τα γειτονικά κράτη ε, συμφωνούν για τη διεξαγωγή ελέγχων σε ε, φορτηγά αυτοκίνητα αλλά πρέπει να παρακολουθούμε τι είδους έλεγχοι έχουν γίνει, με τι συχνότητα και τι αποτελέσματα, πράγμα το οποίο όμως στην πραγματικότητα δεν συμβαίνει ή δεν συμβαίνει συχνά. Εδώ πρέπει η ΕΛΑ λοιπόν να ενισχύσει τη συνεργασία των κρατών μελών και χάρη σε μια ε, ασφαλή βάση δεδομένων και να διευκολύνει το συντονισμό των μέτρων αυτών. Ε, μεταξύ των κρατών μελών. Η καλύτερη υλοποίηση και εφαρμογή της νομοθεσίας του εργατικού δικαίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στους ευρωπαϊκούς δρόμους, είναι βέβαια αρμοδιότητα των κρατών μελών, αλλά όπου υπάρχουν ψηφιακά συστήματα για την ανταλλαγή στοιχείων μεταξύ των αρχών, μπορεί η ΕΛΑ να τα ε, προαγάγει και να τα υποστηρίξει. Ε, επί παραδείγματι, το Ευρωπαϊκό Μητρό Οδικών Μεταφορών, Επιχειρήσεων Οδικών Μεταφορών, ε, είναι ένα πολύ σημαντικό, μια πολύ σημαντική ευκαιρία και έχουμε χάρη σε αυτήν, χάρη σε αυτό το δίκτυο, ένα σύστημα, μια δυνατότητα να παρακολουθούμε την κίνηση των φορτηγών αυτοκινήτων στους ευρωπαϊκούς δρόμους. Μια ευκαιρία που θα πρέπει να αξιοποιήσουμε. Και έτσι είναι εύκολο να διαγνωστεί αν ένας ε, επιχειρηματίας, αν μια επιχείρηση οδικών μεταφορών έχει παραβιάσει στο παρελθόν ή επανειλημμένα τις κοινωνικές διατάξεις. Οι επιθεωρητές εργασίας λοιπόν θα πρέπει να έχουν στη θέση τους τα μέσα εκείνα που θα τους επιτρέπουν να επαληθεύουν τις συνθήκες απασχόλησης των εργαζομένων, των οδηγών δηλαδή των φορτικών αυτοκινήτων, με αποτελεσματικούς ελέγχους των όρων εργασίας που θα εξασφαλίσουν ε, ένα υγιές και δίκαιο σύστημα ε, και σε όρους κοινωνικούς ε, για τις οδικές μεταφορές στην Ευρώπη. Περιμένω τις προτάσεις των συναδέλφων, τα σχόλιά τους, τις επικοδομητικές τροπολογίες και προθεσμία ε, ορίζουμε την Τετάρτη, την επόμενη Τετάρτη 12 του μηνός, στις 12 το μεσημέρι. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία σκιώδη συγγετρία. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είχα ήδη πει ότι δεν μπορώ παρά να υποστηρίξω την πρόταση για αυτή την Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας. Πολλό δε μάλλον που τα αρχικά είναι «έλα», όπως και το δικό μου όνομα. Τώρα έρχομαι στα πιο σοβαρά. Όλες οι ε, δράσεις που στόχο έχουν την εξάλληψη των ε, καταχρήσεων, την καλύτερη συνεργασία μεταξύ των δημόσιων αρχών και των κρατών μελών, την καλύτερη ε, ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ εργατών και εργαζομένων. Όλες αυτές οι πρωτοβουλίες χρήζουν θερμής υποστήριξης, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση εδράζεται στις ελευθερίες ε, κυκλοφορίας εμπορευμάτων ε, και διακίνησης προσώπων. Οπότε και η κινητικότητα των εργαζομένων είναι πολύ σημαντικό θέμα. Θα πρέπει οι εργαζόμενοι να γνωρίζουν ποια είναι τα δικαιώματά τους στο α ή β σύστημα. Αλλά και οι εργοδότες θα πρέπει να γνωρίζουν ποιε είναι οι υποχρεώσεις τους με, στην α ή β ενόμη τάξη. Γι' αυτό και η Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας θα μπορούσε να είναι μια πλατφόρμα στην οποία όλοι οι ενδιαφερόμενοι και οι δύο πλευρές, δηλαδή εργοδότες και εργαζόμενοι, θα βρίσκουν τις ε, πληροφορίες που τους ενδιαφέρουν για τις διατάξεις που ισχύουν στις 28 χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ποιο είναι το σύστημα αμοιβών, ποιες είναι οι διατάξεις για τις συλλογικές διαπραγματεύσεις, ώστε να περιοριστούν οι καταχρήσεις και οι παραβιάσεις. Γιατί τα συστήματα, τα εθνικά συστήματα συλλογικών διαπραγματεύσεων είναι πολύ διαφορετικά. Και μάλιστα στη Γαλλία οι αμοιβέ προσδιορίζονται με βάση πάρα πολλούς διαφορετικούς παράγοντες και συνιστώσεις. Όλες αυτές οι πληροφορίες είναι πολύ χρήσιμες και για τους επιχειρηματίες, ιδιαίτερα τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες που δεν έχουν τη βοήθεια γραφείων ε, νομομαθών για να ε, ξέρουν τι συστήματα ισχύουν. Είναι σημαντικό λοιπόν αυτή η Ευρωπαϊκή Αρχή να λειτουργήσει ω πλατφόρμα ανταλλαγή πληροφοριών και να διαθέτει μια ενημερωμένη βάση δεδομένων που θα είναι μεταφρασμένη σε όλε τι χώρε Ευρωπαϊκή Ένωση για να βοηθήσει του εργοδότε και του εργαζομένου. Είναι πολύ σημαντική και αξιέπαινη αυτή η πρωτοβουλία. Ο συντάκτη, ο κύριος Μιχαήλ Ντέτχεν, τόνισε τον όρο οργανισμό γιατί αρχικά προτάθηκε το γραφείο, Ευρωπαϊκό Γραφείο Εργασίας, η Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας. Χαίρομαι που ο εισηγητής προτείνει να γίνει οργανισμός, Ευρωπαϊκός Οργανισμός Εργασίας. Συμφωνώ με την αλλαγή της ονομασίας, γιατί με τη σύσταση ε, οργανισμών ε, σε τέτοιες περιπτώσεις ε, καλό θα ήταν να έχουμε ε, μία ενιαία διατύπωση και έναν εναρμονισμένο ορισμό. Καλό θα ήταν λοιπόν και αυτή η αρχή να μετονομαστεί σε οργανισμό για να μην έχουμε καμία αμφιβολία για τις αρμοδιότητές της. Τώρα σε ό,τι αφορά την εποπτεία, τον έλεγχο και τη διαμεσολάβηση. Εγώ είμαι υπέρ της ανταλλαγής πληροφοριών, είμαι υπέρ της συνεργασίας, είμαι υπέρ των κοινών ελέγχων υπό τον όρο της Συμφωνίας των Κρατών Μελών να γίνουν τέτοια έλεγχη, αλλά είναι σημαντικό ε, οι ε, ε, δραστηριότητες της, του οργανισμού αυτού να μην σφετερίζεται ούτε εθνικές αρμοδιότητες, ούτε αρμοδιότητες των εθνικών επιθεωρήσεων εργασίας, που αυτές είναι επιφορτισμένες με τον έλεγχο. Ούτε θα πρέπει οι αρμοδιότητες του, της αρχής αυτής να υποκαθιστά άλλες αρμοδιότητες που προκύπτουν από το Ευρωπαϊκό, από το Ενωσιακό Δίκτυο. Επίσης, θα πρέπει να δούμε που θα, ε, που θα στεγαστεί αυτή η νέα αρχή, σε ποια χώρα θα έχει την έδρα της. Ελπίζω όλα αυτά τα σχόλια να ληφθούν υπόψη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με μια πιο ισορροπημένη γεωγραφική κατανομή και επίσης καλό θα ήταν ε, η έδρα που θα επελέξουμε να λάβει υπόψη και το μεγάλο αριθμό μετακινούμενων ε, εργαζομένος στο συγκεκριμένο κράτος μέλος. Σίγουρα δεν θα πρέπει να ε, εμπλακούμε στις αρμοδιότητες ή να μπούμε στα χωράφια των ε, εθνικών επιθεωρήσεων εργασία, αλλά να τι βοηθήσουμε να διευκολύνουμε την ανταλλαγή των πληροφοριών μεταξύ τους και γι' αυτό θα πρέπει να προσδιορίσουμε τις αρμοδιότητες του οργανισμού που θα πρέπει να εξυπηρετεί την ανέβρεση και την ανταλλαγή των κατάλληλων πληροφοριών, αλλά κυρίως θα είναι μια πλατφόρμα για τον περιορισμό των παραβιάσεων κατά την δημιουργία ή πρόσληψη, κατά την ε, μετακίνηση των εργαζομένων, ώστε να αποφευθούν παραβιάσεις ή χρήση ό,τι αφορά τις συλλογικές διαπραγματεύσεις ή τον προσδιορισμό των αμοιβών. Η ομάδα μου το ΕΛΚ θα καταθέσει τροπολογίες ε, για τη γνωμοδότηση αυτή και ευελπιστώ ότι σε συνεργασία με τον συντάκτη και τους υπόλοιπους και θα βρούμε τις καλύτερες συμβαστικές λύσεις. Ευχαριστούμε. Ο κ. Λαδόφσκι από το ECR. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τον ε, κύριο Ντέτχεν για την εκπόνηση του σχεδίου γνωμοδότησης. Δυστυχώς όμως ε, το σχέδιο αυτό δεν έλαβε υπόψη της επιφυλάξεις ε, της ομάδας ECR παρόλο που τις είχαμε διατυπώσει και έχουμε όλο και περισσότερες αφιβολίες για το αυτό το όργανο με τη μορφή που προτείνεται θα ανταποκριθεί ε, στην αποστολή της ενίσχυσης εφαρμογής του ενωσιακού δικαίου. Γιατί παρόλο που δεν, το λέμε, δεν το λέμε οργανισμό, φαίνεται ότι αυτή η Ευρωπαϊκή Αρχή είναι οργανισμός. Πώς προκύπτει αυτή η νέα ορολογία. Γιατί από τη μια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποτίθεται θέλει να περιορίσει τη γραφειοκρατία και από την άλλη δημιουργεί ακόμη έναν οργανισμό που δεν τον λέει οργανισμό, αλλά τα αποτελέσματά του θα είναι παρόμοια με οργανισμό. Σίγουρα ωραίο το όνομα Έλα, είναι και ωραίο πολωνικό όνομα. Αλλά τώρα αν θα είναι οργανισμός, αν θα είναι γραφείο ή αν θα είναι αρχή, δεν μας ενδιαφέρει ε, το θέμα. Είναι τι αρμοδιότητες θα είναι. Πάντως το όνομα είναι ωραίο, συμφωνώ με την κυρία Κουκασιεύσκα. Τώρα, ποια θα είναι οι αρμοδιότητες. Υποτίθεται ότι θα, ε, θα λύσει αποτελεσματικά και τα προβλήματα στον τομέα των μεταφορών η νέα αρχή. Επίσης θα διευκολύνει την καλύτερη συνεργασία και την ενέργεια ελέγχων ε, μεταξύ των κρατών μελών στα πλαίσια του Eurocontrol. Βέβαια, μόνο στην αιτιολογική σκέψη αναφέρεται κάτι τέτοιο. Στα πλαίσια της συνεργασίας ε, στην Eurocontrol είχαμε πολύ γλωσσο λεξικό, λεξιλόγια προκειμένου να διευκολυνθεί η συνεργασία μεταξύ των ελεκτικών χωρών και επίσης ε, πολύ γλωσ... έντυπο, έντυπο δηλαδή σε πολλές γλώσσες για να διευκολυνθεί ο έλεγχος και η συνεργασία μα αυτή η συνεργασία ήδη υπάρχει στην Eurocontrol και είναι αποτελεσματική. Δεν χρειαζόμαστε ένα επιπλέον γραφειοκρατικό οργανισμό. Ούτε η πρώτη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ούτε η γνωμοδότηση δείχνει πραγματικού τρόπου υποστήριξη των επιχειρήσεων. Γιατί αυτό είναι σημαντικό. Πώς θα βοηθήσουμε τους επιχειρηματίες και επίσης τι θα γίνει με την απόσπαση των εργαζομένων. Το έργο της Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας θα πρέπει να είναι κυρίως ε, ενημερωτικό, πληροφοριακό, ε, πληροφόρησης και των εργοδοτών και των εργαζομένων. Τώρα, σε ό,τι αφορά τους εργοδότες, Μόνο η τροπολογία 2 αναφέρεται στις καταχρήσεις που γίνονται από τις μεταφορικές εταιρείες. Σε πολλές περιπτώσεις ε, γίνεται πολύ ευρία παρουσίαση των αρμοδιοτήτων, είναι πολύ ε, γενική αναφορά των αρμοδιοτήτων και τα άρθρα 2 και 5 ε, αμφιβάλλω αν ε, ε συμβιβάζονται με, την, με το άρθρο 344 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, φαίνεται ότι μερικές φορές η, αρχή θα κάνει διαμεσολάβηση μεταξύ των κρατών μελών ή θα διευκολύνει το συντονισμό ή τη διενέργεια των κοινών ελέγχων. Ε, Στι τροπολογίες 14 και 18... Ε, χορηγούν στη νέα αρχή αρμοδιότητες που εμφανώς σφετερίζονται εθνικές ελεκτικές αρμοδιότητες το σχέδιο της γνωμοδότησης ε, δυστυχώς όχι μόνο δεν διόρθωσε τις αδυναμίες της πρώτης Ευρωπαϊκής ε, Επιτροπής, αλλά δημιούργησε και κάποια σύγκρουση αρμοδιοτήτων με τις εθνικές αρμοδιότητες και τις αρμοδιότητες των εθνικών επιθεωρήσεων εργασίας. Φαίνεται ότι το γραφείο αυτό όχι απλώς συντονίζει ελέγχους, αλλά ε, διενεργεί ελέγχους, έχει διαμεσολαβητικό ρόλο ή ξεκινά διαδικασίες επί παραβάση των υποχρεώσεων των κρατών μελών. Φυσικά και θα καταθέσουμε ως ECR τροπολογίες για την γνωμοδότηση, αν και γενικώ έχουμε αρνητική διάθεση απέναντι στη γνωμοδότηση. Και μάλιστα μετά την παρουσίαση είναι ακόμη πιο αρνητική η εντύπωσή μας. Παρ' όλα αυτά θα καταθέσουμε τροπολογίες επιχειρώντας να βελτιώσουμε κάπως τη γνωμοδότηση του κ. Ευχαριστώ ε, κύριε Ζωτόφσκι. Ο κύριος Ράντος από τους φιλελεύθερους έχει να πει κάτι. Ο κύριος Ράντος από τους φιλελεύθερους έχει να πει κάτι. Όχι. Οπότε ο κύριος Μπαχ. Oui, merci, Ευχαριστώ, Ντομινίκ. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να συγχαρώ τον Μίχαελ Ντέτσιν για τη δουλειά του. Όταν ανέφερε την ενιαία αγορά και τις δίκαιες συνθήκες, θεμητές συνθήκες, ε, έθιξε ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα και γι' αυτό θεωρώ ότι η ίδρυση ενό ε, οργανισμού ή μια αρχής, όπως το πούμε, πρέπει να έχει και τα κατάλληλα... Πρέπει να συνοδεύεται και από τα κατάλληλα κονδύλια, ώστε μπορεί να κάνει σωστά τη δουλειά του. Οπωσδήποτε είναι κατεπίγουσα η ίδρυσή του οργανισμού. Η ιδέα δεν είναι καινούρια. Ο Μισελ Μπαρνιέ το 2013, όταν ήταν ακόμα επίτροπος για την εσωτερική αγορά, είχε ε, προτείνει μια τέτοια ιδέα. Είναι ακόμα πολύ σημαντικότερο βέβαια τώρα που έχουν προκύψει πολλές νέες και αθέμητες μορφές ε, απασχόλησης ο ρόλος μας δεν θα είναι βεβαίως τόσο πολύ εδώ να παρακολουθήσουμε την ίδρυση του κανονισμού όσο στην Επιτροπή Απασχόλησης, αλλά πρέπει να έχει την ε, αρμοδιότητα να εξετάζει και ζητήματα της απόσπασης. Ως προς τις αρμοδιότητες συγκεκριμένα του οργανισμού φοβούμε ότι εάν δεν υπάρξουν επαρκή μέσα για την ε, επίτευξη του έργου του οργανισμού αυτού κινδυνεύει να μείνει μόνο στο χαρτί ή απλώς ε, να είναι ένας τίγρης ξεδοντιάρης αυτός ο οργανισμός. Ε, θα πρέπει να ετοιμάζει μια έκθεση κάθε χρόνο για τους ελέγχους που έχουν υλοποιηθεί, για τις ε, συνέπειες που προτείνονται έτσι θα πρέπει να υποστηριχθεί, αλλά βλέπουμε ότι υπάρχουν κράτη που δεν υποστηρίζουν, δεν υπάρχει καν απαρτία σε επίπεδο κρατών για να υποστηριχθεί αυτή η αρμοδιότητα και θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και αυτό δίνω ένα μόνο παράδειγμα, να προσφέρει τα κατάλληλα μέσα στον οργανισμό. Σημείο κρίσιμο για μένα, άλλωστε το ανέφερε και η κυρία Λουκασέφτσκα, η συνάδελφος, Κρίσιμο σημείο λοιπόν θα είναι το πώς μπορεί να υλοποιηθεί η συνεργασία με τα κράτη-μέλη. Από εκεί θα προκύψει η στη θέμενη αξία του φορέα αυτού. ο οποίος θα πρέπει να περιορίζεται μόνο στην επανάληψη των αρμοδιοτήτων των κρατών μελών, αλλά να έχει προστιθέμενη αξία, να δρά κατά τρόπο διαμεσολαβητικό ε, σε περίπτωση ε, διαφορών σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, αλλά πάνω απ' όλα να προλαβαίνει την ανάδειξη των διαφορών και προσφυγών στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο διαμεσολαβώντας στον τρόπο με τον οποίο τα κράτη βλέπουν ε, τα ζητήματα των αρμοδιοτήτων αυτών. Και η συνεργασία των κοινωνικών εταίρων θα έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία για να επιτύχει ο οργανισμός αυτό στο έργο του. Θα πρέπει δηλαδή οι κοινωνικοί εταίροι να συμμετέχουν και όχι μόνο συμβουλευτικά εκ των υστέρων, αλλά εξ αρχής και με πολύ ε, δραστήριο τρόπο, για να μην πω προδραστικό, ε, να συμμετέχουν στη διαμόρφωση και το έργο του οργανισμού αυτού. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Το σχέδιο γνωμοδότησης του Μισελ πάει προς τη σωστή κατεύθυνση και προσθέτει πολλά στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τώρα να συμπληρωθεί με τον κανονισμό των υπηρεσιών αυτών είναι κάτι το οποίο προσθέτει στις αρμοδιότητες του οργανισμού. Η ευρωπαϊκή αυτή αρχή πρέπει να ελέγχει τις καταχρηστικές πρακτικές όταν ε, υπάρχουν περίδιες προσλήψεις και θα πρέπει να φροντίζει και οι κοινωνικές ε, παροχές να δίνονται έτσι όπως πρέπει και όχι μόνο μόνος στόχος να είναι η μείωση του κόστους εργασίας. Πρέπει να επεκταθούν οι αρμοδιότητες και στην καταπολέμηση της ψεύτο αυτόνομης εργασίας. Στηρίζω επίσης τις τροπολογίες που έχουν σαν στόχο να συμπεριληφθούν στις αρμοδιότητες της αρχές η πρόσφαση σε πραγματικό χρόνο στα στοιχεία των ε, επιχειρήσεων μεταφορών που δρούν στην Ευρώπη. Πρέπει να είναι δυνατόν να υπάρχει αυτός ο έλεγχος στους δρόμους. Όμως πιστεύω ότι μπορούμε να πάμε και πιο μακριά στα προνόμια της αρχής αυτής να μπορεί να συνεργαστεί με εθνικέ αρχέ ή να μπορεί να παρέμβει όταν υπάρχει σύγκρουση ανάμεσα σε δύο εθνικέ αρχέ. Δεν πρέπει να είναι μόνο διαμεσολαβητή, αλλά θα πρέπει να μπορεί και να αποτελέσει τον διαιτητή και να λαμβάνει και δεσμευτικέ αποφάσει. Ε, χαίρομαι και ελπίζω θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε την ανταλλαγή απόψεων με τον εισηγητή. Η κυρία Αρνοτού. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και εγώ τον εισηγητή. Ξέρετε, ο Ζώσο Κλεμονσό είχε πει ότι αν θέλετε να θάψετε ένα πρόβλημα, δεν έχετε παρά μια επιτροπή. Ε, νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο εξακολουθεί να ισχύει έναν αιώνα αργότερα. Γιατί όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται αντιμέτωπη με τα όρια τη τελικά, τι κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, βγάζει από το καπέλο μια νέα, ένα νέο οργανισμό. Πάλι για να έρθω στον Κλεμοσό, τελικά ε, όταν υπάρχει πρόβλημα ε, ξαφνικά υπάρχει μεγάλη γονιμότητα και εμφανίζονται καινούρια στοιχεία. Εδώ δεν μπορεί να νομίζουμε ότι μόνο και περισσότεροι Ευρώπη θα λυθούν τα προβλήματα, γιατί στο κάτω-κάτω ο κόσμος το πιστεύει όλο και λιγότερο. Καλά θα κάνει η Επιτροπή να εφαρμόσει το είδη ήδη ισχύουν και να ε, αποφεύγει τις καταχρήσεις. Πιστεύετε όμως ότι με την νέα αυτή αρχή θα βελτιωθεί η κατάσταση που ζουν οι πολίτες μας με τη δουλειά τους, με τόση ανεργία που πλήττει την Ευρώπη. Εγώ πιστεύω ότι η αρχή αυτή θα είναι ανίκανη όπως είναι και οι εθνικές αρχές γιατί αυτό που φταίει είναι η ίδια η αρχή στην οποία βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι αυτό το σύστημα το οποίο έχει δημιουργήσει ένα δόγμα τεράστιου ανταγωνισμού. Έτσι λοιπόν αυτές οι υπερβολικές ε, ρυθμίσεις πιστεύουμε ότι είναι ανεύθυνες, άσε που δεν ε, μπορούν καν ε, να τηρηθούν, δεν είναι ρεαλιστικές. Αυτό που έχει γίνει με τις μέχρι τώρα ρυθμίσεις είναι ότι έχουμε άκρατο ανταγωνισμό, από το οποίο πλήττονται οι εργάτες μας, οι μεταφορείς μας και βέβαια έχουμε και τους μισθούς οι οποίοι έχουν πέσει κατά πολύ από τους φτηνούς εργαζόμενους που εισάγουμε. Όπως καταλαβαίνετε, είμαι ιδιαίτερα επιφυλακτική για αυτήν την πρόταση, παρόλο που λέει ότι θα είναι ένα μεγάλο βήμα προς την κοινωνική Ευρώπη. Ίσως να υπάρχουν καλές προθέσεις, αλλά οι καλύτερες προθέσεις του κόσμου οδηγούν στην ε, κόλαση, γιατί και η κόλαση είναι γεμάτη καλές προθέσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Τώρα θα δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή από τη Γενική Διαθέση MOVE. Παρακαλώ. ποιο, Εσείς. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Καλημέρα σε όλους. Πρώτα απ' όλα, σας ε, ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον εισηγητή και ευχαριστώ και για την στήριξή σας για τη δημιουργία της αρχής αυτής και προκειμένου να συμπεριληφθεί στις δραστηριότητε της αρχής και το θέμα των μεταφορών. Θα είμαι σύντομος, θα περιορίσω την παρέμβασή μου σε τέσσερις παρατηρήσεις. Πρώτον, σημειώνω τις τροπολογίες του εισηγητή για να ενισχυθεί η υποχρέωση των χωρών μελών να συνεργάζονται με την αρχή αυτή. Ε, προθεσμία προκειμένου οι χώρες μέλη να δίνουν πληροφορίες. Και αν δεν υπάρχει συνεργασία των χωρών μελών, τότε θα πρέπει να ενημερώνεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που θα παίρνει τα κατάλληλα μέτρα. Η τροπολογία αυτή ευθυγραμμίζεται με πολλές παρεμβάσεις που έγιναν από τους ευρωβουλευτές της Επιτροπής αυτής όταν για πρώτη φορά είχαμε παρουσιάσει την πρότασή μας. Δεύτερη παρατήρηση. Σημειώνω ότι ο εισηγητής θέλει να επικεντρωθεί στη, στο peer reviews, ε, τις αξιολογίες μεταξύ ομοτήμων και την ανταλλαγή απόψεων μεταξύ αντίστοιχων αρχών. Τρίτον, σημειώνουμε επίσης ότι ο συγητής προτείνει να συμπεριλάβουμε και μνήα και στις οδικές μεταφορές και στις ενέργειες μεταφορές βάσει του κανονισμού του 2008. Πράγματι, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην πρότασή της επικεντρώνεται στις οδικές μεταφορές και πιστεύω ότι όντως υπάρχει επίγουσα ανάγκη να βελτιωθεί η εφαρμογή, η τήρηση των κανόνων εδώ. Δεν υπάρχει η καμία υπηρεσία στις οδικές ε, μεταφορές ή τις ενέργειες, πέρα από την Ιάσα. Οπότε εδώ θα μπορούσε να υπάρχει κάποια επέκταση των αρμοδιοτήτων της ΕΑΣΑ. Η μελλοντική αρχή πάντως δεν έχει έναν ε, περιορισμένο κλειστό κατάλογο αρμοδιοτήτων. Θα μπορούσαν να επεκταθούν οι αρμοδιότητες αυτές και στις οδικές μεταφορές αλλά και στις ενέργειες. Μιλάμε πολύ για τις ενέργειες μεταφορές. Όπως είπε και ο Ρίκολο, λέει ο Γενικός μου Διευθυντής, η Γενική Διευθυνσή μου ετοιμάζει έκθεση για τις κοινωνικές επιπτώσεις στην ε, αεροπορία που θα είναι έτοιμη σύντομα. κοιτάμε έτσι να δούμε αν χρειάζεται ένας νέος μηχανισμός ε, τήρησης ή κάποια επέκταση των, αρμοδιοτήτων της ΙΑΣΑ. Οπότε μένει ανοιχτό αυτό το ζήτημα. Και η τελευταία μου παρατήρηση έχει να κάνει με την τροπολογία 16 όπου προτείνει ο εισηγητής οι επιθεωρητές να έχουν απευθείας πρόσβαση στις πληροφορίες του EMI. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στηρίζει απόλυτα τον στόχο αυτό της απευθείας πρόσβασης στην ενημέρωση της πληροφορίας των επιθεωρητών. Το ερώτημα είναι κατά πόσο ο ιδρυτικός κανονισμός της ευρωπαϊκής αυτής αρχής είναι και ο κατάλληλος χώρος για να τεθεί αυτή η διάταξη. Και αυτό είναι που θέλουν, οι, που αναρωτιούνται και τρεις εισηγητές του πακέτου. Αυτές είναι οι τέσσερις παρατηρήσεις μου. Και για κάτι που είπε ο κύριος Λοτόφσκι, ο οποίος έφυγε. Αλλά ποια είναι η αξία για τις επιχειρήσεις η δημιουργία μιας τέτοιας αρχής. Εγώ πιστεύω ότι η απάντηση είναι απλή. Οι επιχειρήσεις που συμμορφώνονται με τους ευρωπαϊκούς κανόνες έχουν πλεονέκτημα απέναντι στις άλλες που δεν συμμορφώνονται και που σε αυτές θα επιβάλλονται κυρώσεις εφόσον δεν συμμορφώνονται από την ε, νέα αυτή αρχή. Και για τον κύριο Μπαχ, για το σαφή ρόλο των συνδικάτων. Πράγματι, από ό,τι έχω καταλάβει, προβλέπει στη δομή του σχεδίου κανονισμού ότι θα έχουν ρόλο τα συνδικάτα στην ομάδα των stakeholders, όπως λέγονται. Αυτά είχα να πω, αλλά όπως είπα και στην αρχή, υπάρχει μια διατραθετική εκτίμηση απέναντι στην νέα αυτή αρχή. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Θα δώσω το λόγο στον εισηγητή μας τώρα για να καταλήξει. Ευχαριστώ πολύ. Καταγράφω λοιπόν τις παρατηρήσεις ως ε, προσθήκες και ευχαριστώ πολύ κυρία Λουκασιέτσκα παραδείγματι πέραν σημειολογικών ζητημάτων που θα έχουμε την ευκαιρία να διευκρινίσουμε νομίζω ότι ως προς την ουσία συμφωνούμε σε μεγάλο βαθμό. Για τον κύριο Μπάχ επίσης, τον οποίο και ευχαριστώ για την ε, πρόταση για πιο ε, στενή συνεργασία των κοινωνικών εταίρων. Πιστεύω ότι έχοντας και αντίστοιχη εμπειρία από τη χώρα προελεύσεως μπορούμε να ε, αξιολογήσουμε θετικά τη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων. Αυτά και θα ήθελα και άλλες τροπολογίες να δω. Περιμένω βεβαίως τη συνεργασία με τους συναδέλφους. Μάλιστα. Ευχαριστούμε κύριε Τέτια. Να σας υπενθυμίσω ότι η για την κατάθεση προτροπολογιών λίγη στις 12 Σεπτεμβρίου για να ψηφίσουμε στην Επιτροπή μας στις 9 Οκτωβρίου. Περνάμε τώρα στο τρίτο θέμα της απογευματινής ημερήσιας διάταξης, στα πρότυπα επιδόσεων για τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα των νέων βαρέων επαγγελματικών οχημάτων. Πρόκειται για γνωμοδότηση που θα χορηγήσουμε στην αρμόδια κατουσία επιτροπή που είναι η ΕΜΒΗ, Επιτροπή Περιβάλλοντο. Η κυρία Βιρκούνεν, ε, κανονικά είναι η συντάκτρια τη γνωμοδότηση. Ε, είναι εδώ η. Και να προ... Έφυγε με μια ταλίκα, λέει ο κύριο Βαντερκάμπ. Άλλο από την αναπληρώνει. Μας έφυγε η συγγήτρια.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 Ο κύριος Βαντενκάμπ. Θα την αντικαταστήσετε εσείς. Ωραία. Ο κύριος Βαντενκάμπ έχει το λόγο που αναπληρώνει την ε, εισηγήτρια, την κυρία Βίρκουναν. Συγγνώμη, πρόεδρε, το έχω ξεχάσει ότι έπρεπε να αντικαταστήσω την ε, κυρία Βίρκουναν. Θα σας διαβάσω λοιπόν τι μου έδωσε, τι μου εμπιστεύτηκε. Η... Και θα... Πώς στα αγγλικά. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε τις ίδιες μειώσεις ε, διοξιδίου του άνθρακα για τα βαρέα επαγγελματικά οχήματα, όπως προτείνει και για τα επιβατικά και για τα φορτηγά, φορτηγάκια. Δηλαδή το 2025, 15% μείωση και για το 2030 30% μείωση και για τα βαρέα επαγγελματικά οχήματα. Η στόχη αυτή, κατά τη γνώμη της ηγήτρης κυρίας Βερκούνεν, είναι πολύ φιλόδοξη για τα βαρέα επαγγελματικά οχήματα, μια και δεν μπορούμε να συγκρίνουμε τα οχήματα αυτά με τα επιβατικά ή τα μικρά φορτηγά. Η επίτευξη αυτής της μείωσης ε, θα γίνει μόνο αν συνδυαστούν κάποιες λύσεις. Επίσης, οι μειώσεις εκπομπών ε, μπορούν να επιτευχθούν με την ανάπτυξη λύσεων, όπως ε, βελτιστοποίηση του φορτίου, πλατούνινγκ, βοήθεια στους οδηγούς, ε, κατάρτιση των οδηγών, δημιουργία εναυσμάτων για την αναβάθμιση του στόλου χυμάτων, η εξασφάλιση επενδύσεων στις υποδομές, την ανάπτυξη και τη συντήρηση. Κάτι που είναι πολύ σημαντικό είναι η ουδετερότητα τεχνολογική. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη λοιπόν όλες τις καινοτομίες. Δυστυχώς όμως ε, η πρόταση με τον τρόπο υπολογισμού που περιέχει αυτή τη στιγμή δεν είναι τεχνολογικά ουδέτερη. Εξού και η συγγετρία προτείνει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να θεσπίσει υπολογισμούς από το φρέος στον τροχό, well to will και να θεσπίσει αυτόν τον τρόπο υπολογισμού μέχρι το 2022 ε, αντικαθιστώντας την παρούσα μέθοδο δεξαμενή προς τροχό, tank to wheel, και να λάβει υπόψη ε, και την τελική χρήση των οχημάτων καθώς και τις νέες τεχνολογίες. Θα πρέπει να βρούμε σωστή ισορροπία μεταξύ του στόχου, της πρόθεση της καινοτομίας και την ενίσχυση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας σε συνδυασμό με τη δημιουργία ε, εξειδικεύσεων ε, θέσεων μάλλον θέσεις απασχόλησης. Πολλά χαιρετίσματα από την Χένα. Βιρκούνεν. Ευχαριστούμε και ευχαριστώ που έσωψες να αναπληρώσεις τελευταία στιγμή την ε, εισηγήτρια. Περνάμε στους και ηγητέ. Η κυρία Ρεβόντα Λόν από τους σοσιαλιστές. Παρακαλώ. Ε, τα πρότυπα εκπομπών για τα ελαφρά ε, οχήματα υπάρχουν εδώ και καιρό. Για τα βαρέα όμω επαγγελματικά οχήματα πρώτη φορά έχουμε τέτοια πρότυπα εκπομπών. Επιτέλου, χαιρόμαστε ιδιαίτερω. Θα πρέπει να ανταποκριθούμε στι κλιματικέ προκλήσει και να σταθούμε στο ύψο των περιστάσεων. Γιατί αν θέλουμε να σεβαστούμε τι δεσμεύσει του 2050 που έχουμε λάβει στη Συμφωνία των Παρισίων, θα πρέπει από τώρα να δράσουμε και όσο θα βλέπουμε τις συνέπειες των κλιματικών αλλαγών θα είναι ήδη πολύ αργά. Η αυτοκινητοβιομηχανία είναι από του προμαχώνες της ευρωπαϊκή οικονομίας. Κάτι που ισχύει όμως για τα ελαφρά οχήματα θα πρέπει να ισχύει και για τα βαρέα επαγγελματικά οχήματα, παρόλο που δεν βρίσκονται στο επίκεντρο της ε, δημόσιας προσοχής. Γι' αυτό θα πρέπει να ετοιμάσουμε τις ε, καινοτομίε και στον κλάδο αυτό. Κάτι που είναι προ και της ανταγωνιστικότητάς μα αλλά και του πλανήτη μα. Βέβαια, όταν λέμε επαγγελματικά, βαρέα επαγγελματικά οχήματα, έχουμε πολλέ χρήσει, πολλά είδη οχημάτων, ένα πολυσύνθετο τοπίο και διαφορετικέ χρήσει. Μερικά οχήματα θα διανύσουν ένα εκατομμύριο χιλιόμετρα καθ' όλη τη διάρκεια τη ζωή. Μήπω μπορείτε να μιλάτε λίγο πιο σιγά, κύριε Βαντερκάμπ. Ένα εκατομμύριο χιλιόμετρα λοιπόν θα διανύσουν μερικά τέτοια βαρέα επαγγελματικά οχήματα, ενώ άλλα θα κάνουν καθημερινά 18 ώρα ταξίδια μεταφορά επιβατών. Ε, δεν έχουμε όμως αρκετή απόσταση για να αξιολογήσουμε τι είναι πραγματικά εφικτό σήμερα. Γι' αυτό θα πρέπει σε μια πρώτη φάση να έχουμε διαφοροποιημένες προσεγγίσεις, ώστε να υιοθετήσουμε όπου είναι εφικτό τον χρήσιμο ρυθμό. Η αναθεώρηση που προτείνεται για το 2022 θα είναι σημαντικό ορόσημο για να τελειοποιήσουμε την νομοθεσία, να καλύψουμε περισσότερα οχήματα και ενδεχομένω ε, να υιοθετήσουμε πιο φιλόδοξου στόχου. Γιατί όλοι οι κλάδοι θα πρέπει να συμβάλλουν στην καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών και θα πρέπει να εξαιρούνται οι οδικέ μεταφορέ. Δεν έχουμε καμία έτοιμη τεχνολογική λύση θα πρέπει να μειώσουμε περαιτέρω τι εκπομπέ, θα χρειαστεί όμω χρόνο. Επίση, να εκμεταλλευτούμε τι νέε τεχνολογίε, γιατί όλε έχουν πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Υπάρχουν πάντω πολλέ ελπιδοφόρε ενδείξει από τα ανανεώσιμα καύσιμα ανάλογα και με τις αγορές. Θέλουμε λοιπόν μια σωστή αφετηρία ώστε στο μέλλον να εμπεδώσουμε, να εδραιώσουμε την ομοθεσία μας και θα πρέπει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να φανεί πιο φιλόδοξο την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε όλα αυτά τα θέματα. Σας ευχαριστούμε κυρία Λεβόνταλόν. Ο κύριος Ράντος από τους Φιλελεύθερους. Γιώζο, έχει το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Εκ μέρους των Φιλελευθέρων θα ήθελα να στηρίξω την γνωμοδότηση που αποκρίνεται στις σύγχρονες βιομηχανικές και περιβαλλοντικές πολιτικές Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άλλωστε η πρόταση αυτή είναι παρόμοια με τη γνωμοδότηση για τις εκπομπές ε, των επιβατικών αυτοκινήτων, των επιβατικών οχημάτων. Ε, και είναι σημαντικό να έχουμε πρότυπα αντίστοιχα και για τα βαρέα επαγγελματικά οχήματα. Γι' αυτό και η θέση των φιλελευθέρων είναι η ίδια με αυτή για τα επιβατικά οχήματα. Είμαστε υπέρ της μείωσης των εκπομπών, ε, όπως προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και για τα βαρέα επαγγελματικά οχήματα και είμαστε διαλλακτικοί και προς πιο φιλόδοξες προσεγγίσεις. Επίσης, ε, η παραγωγή επικαλούμενη Κάποιες επιστημονικές μελέτες ε, θεωρούν ότι η μειώση κατά 15 και 30% μέχρι το 2030 είναι υπερβολικά φιλόδοξη και η σύγχρονη τεχνολογική πρόοδος δεν επιτρέπει την υλοποίηση αυτών των φιλόδοξων ε, μειώσεων. Άλλωστε, η αναθεώρηση που αναμένεται για το 2022 παρά είναι ε, σε σύντομο χρονικό διάστημα. Δεν θα έχουμε αρκετή απόσταση ε, μετά από δύο-τρία χρόνια. Είναι δυνατόν να αλλάξει τόσο όρεξη και έλευθε η τεχνολογία μέσα σε δύο-τρία χρόνια για να μπορέσουμε να κάνουμε την αναθεώρηση. Πάντως είμαστε υπέρ της πρότασης ε, της ηγήτριας μέχρι το 2022 να αναπτυχθεί η τεχνολογία μέτρηση των εκπομπών, ε, η από την αρχή, από το φρέαρ στον τροχό, well to wheel, γιατί αυτό είναι, αυτό, είναι, αυτό δίνει πραγματικές ενδείξεις ε, για τις πραγματικές εκπομπές. Επίσης, ε, η δεκτοπροσωμείωση, η των οχημάτων ε, σήμερα δεν καλύπτει τις νέες τεχνολογίες. Ε, οπότε, ίσως δεν είναι καλή μέθοδος γιατί δεν καλύπτει ούτε τις τρέχουσες τεχνολογίες ούτε σίγουρα θα καλύψει τις νέες τεχνολογίες που στο μεταξύ θα αναπτυχθούν ε, κατά την προσπάθεια μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Συμφωνώ λοιπόν με την πρόταση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ανανεώσει και να επικαιροποιήσει τις μεθόδους αυτών των προσωμιώσεων που προτείνει, ώστε αυτός, αυτή η μεθοδολογία να γίνει όσο πιο ακριβής γίνεται. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Εκ μέρους των Πρασίνων, τώρα, κύριο Σταλούτ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είναι ένα θέμα που επήγει, γιατί όταν δεν υπάρχει φιλόδοξη πολιτική από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακος, καταλαβαίνετε ότι δεν προχωράμε. Είπαμε ότι θα έπρεπε να μειωθούν κατά 9% οι εκπομπές. Οι χώρες μέλη όμως δεν πετυχαίνουν τους στόχους τους και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε βάλει 40% και στην Ενεργειακή Ένωση. Παρά λοιπόν τις τεχνολογίες που υπάρχουν προκειμένου να μειωθούν οι εκπομπές, αυτό δεν γίνεται. Οι μεταφορείς, οι πελάτες τους δεν τα καταφέρνουν. Τρίτο πρόβλημα. Στις Ηνωμένε Πολιτείε, στην Κίνα και αλλού, όσοι κατασκευάζουν οχήματα ΣΑΒ έχουν φροντίσει για τη μείωση εκπομπών. Εδώ όμως στην Ευρώπη δεν έχουμε τέτοια προγράμματα δράσης, κάτι το οποίο όμως έχει και σαν αποτέλεσμα να πλήττεται η ανταγωνιστικότητά μας. Σύμφωνα με την ε, εξέταση αντικτύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Μόλι τι μεθόδου μπορούμε να έχουμε 15 με 20% μείωση μέχρι το 2025, χωρί καν να λάβουμε υπόψη μας όλες τις παραμέτρους. Η έκθεση αντικτύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής λέει ότι ο στόχος μείον 20% είναι αυτός από τον οποίο θα αποφελθεί περισσότερο κοινωνία μέχρι το 2025, ότι είναι και ένας ρεαλιστικός στόχος και μας εκπλήσει που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν λαμβάνει υπόψη τις συστάσεις της δικιάς της της έκθεσης δικτύπου. Ε, Ευτυχώ που υπάρχουν και πράσινοι. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επίση στην έκθεση αντικτύπου λέει ότι μόνο αν υπάρξει μείωση εκπομπών θα μπορέσει να αυξηθεί και να ισχυθεί η ανταγωνιστικότητα και εμείς θα υποβάλουμε τροπολογίες προς αυτή την κατεύθυνση. Ευχαριστώ. Η κυρία Γκονζάλες Πένιας, εκ μέρους της ΚΟΕ, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, και ευχαριστώ και την κυρία Πινακούνεν για το έργο της. Γνωρίζουμε ότι εδώ και χρόνια στις οδικές μεταφορές έχουμε πολλά προβλήματα. Είναι πρώτα απ' όλα οι σκληρές συνθήκε εργασίας, ο ανταγωνισμός και κανονισμοί όπως αυτός που συζητάμε τώρα που θα έπρεπε να διορθωθεί. Αυτή η σκέψη ότι τα νέα οχήματα θα ρηπαίνουν λιγότερο στο μέλλον είναι ένας καλός τρόπος για να καταπολεμηθούν οι κλιματικές αλλαγές και να ε, μπορέσουμε να τηρήσουμε τους στόχους της Συμφωνίας των Παρισίων. Φυσικά και συμφωνούμε με την πρόθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σταδιακά, αλλά ίσως δεν υπάρχει αρκετή φιλοδοξία όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής, που είναι μόνο τα οχήματα τα οποία παίρνουν περισσότερο. Είναι σημαντικό ο κανονισμός να προχωρήσει, οπότε ίσως δεν γίνεται να βάλουμε σαν πεδίο εφαρμογή τα πάντα, αλλά αν μη τι άλλο εμείς θα υποβάλουμε τροπολογίες έτσι ώστε να μην τεθούν σε κίνδυνο οι στόχοι μείωσης των εκπομπών. Από την άλλη θεωρούμε ότι είναι σημαντικό και θα στηρίξουμε οποιαδήποτε πρωτοβουλία στην Ευρώπη, όπως γίνεται σε άλλες χώρες, η Ιαπωνία, οι Ηνωμένε Πολιτείε, για υποχρεωτικά ελάχιστα επίπεδα για ε, όσους κατασκευάζουν οχήματα, να είναι είτε με ε, μηδενικές εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα ή πολύ χαμηλές. Και να λάβουμε υπόψη μας και τις επενδύσεις και την γρήγορη εξέλιξη νέας γενιάς τέτοιων βαρέων οχημάτων. Το τελευταίο που θέλω να υπογραμμίσω ο ήθιστη είναι ότι το πρόβλημα αυτό μπορεί κανείς να το αντιμετωπίσει από πολλές πλευρές. Σίγουρα πρέπει να δώσουμε περισσότερη βάση στις ε, δημόσιες μεταφορές, στις μαζικές μεταφορές, ε, το τρένο που ρηπαίνει λιγότερο. και σίγουρα και τα οχήματα που ρηπαίνουν λιγότερο. Τις τροπολογίες μας θα τις υποβάλουμε όπως σας είπα και είμαστε αισιόδοξοι. Ελπίζουμε να καταφέρουμε να φτάσουμε σε μια καλή συμφωνία. Πρόεδρο, σε ευχαριστούμε πολύ. Το λόγο έχει τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο κύριος Φιτσκέρα, μέρος της Επιτροπής, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ που προσκαλέσατε την Επιτροπή που μας κάλεσατε να σχολιάσουμε και ευχαριστώ και την εισηγητρή. Είναι σύντομη η έκθεση. Εύκολο να τη σχολιάσουμε. Ένα-δύο πράγματα όμω πρέπει να πω εξ υπαρχή. Καταρχά, εκ μέρου τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλουμε να τονίσουμε πω στόχο μα είναι να αντιμετωπίσουμε ταυτόχρονα τρία ζητήματα. Αφενό, με περιβαλλοντικό, εκπομπέ του άνθρακα δηλαδή που αναφέρθηκαν, Δεύτερον, και είναι πολύ σημαντικό, ε, οι επιχειρήσεις μεταφορών που θέλουμε να κερδίσουν χάρη σε αυτή την ε, πρόταση και αν κοιτάξουμε την μελέτη δικτύπου με την εξοικονόμηση σε όρους καυσίμων κερδίζουν, ε, εξοικονομούν 25.000 ευρώ τα πέντε πρώτα χρόνια από καύσιμα οι επιχειρήσεις μεταφορών. Είναι τεράστιο το ποσό. Είναι ένα τεράστιο κέρδος στους δρόμους στη διάθεσή μας εφόσον υιοθετηθεί η πρόταση και ελπίζουμε ότι θα υιοθετηθεί μέσα στον χρόνο. Τρίτον, επίσης αναφέρθηκε, η ευρωπαϊκή βιομηχανία πρέπει να παραμείνει ανταγωνιστική σε διεθνές επίπεδο. Έχει γίνει και μια παραπομπή σε άλλες ε, ε, δικαιοδοσίες. Κίνα, Ιαπωνία, Ινδία, Ηνωμένε Πολιτείε που ήδη έχουν προδιαγραφές για τα βαρέα οχήματα, πράγμα το οποίο αποτελεί ένα επιπλέον κίνητρο για την παραγωγή νέων τεχνολογιών. Πρέπει λοιπόν να εξασφαλίσουμε πως η δική μας η βιομηχανία θα είναι σε θέση να προχωρήσει και να μην χάσει την, ε, να μην απολέσει την ε, πρωτοκαθεδρία που έχει σε τεχνολογικό επίπεδο. Η προσέγγιση, και νομίζω επισημάνθηκε παρελειμμένος εδώ, είναι σταδιακή. Πρώτη φορά αναλαμβάνουμε πρωτοβουλία ε, ρύθμισης των καυσίμων και άρα έχουμε περιορισμένο πεδίο ως προς τις γνώσεις που διαθέτουμε. Ε, θα θέλαμε βεβαίως όλα τα μεγάλα οχήματα, τα φορτηγά, τα λεωφορεία, ε, τα φορτηγά ε, σύντομης μίσθωσης να μπορούσαμε να τα περιλάβουμε, που μπορεί να είναι διαφορετικές κατηγορίες, αλλά λίγο πολύ έχουν κοινά χαρακτηριστικά, ορισμένα μεταξύ τους, ενώ κάποια άλλα έχουν τελείως διαφορετικά. Ε, είναι τελείως διαφορετικά. Γι' αυτό λοιπόν θέλουμε μια σταδιακή ανάλυση να αναπτύξουμε για τα μεγάλα φορτηγά που καλύπτουν το 75% των, καυσί, των εκπομπών των προερχομένων από φορτηγά. Και γι' αυτό αντιμετωπίζουμε πρώτα αυτά και το 2022 με την αναθεώρηση πιστεύουμε θα μπορέσουμε να καλύψουμε και τα λοιπά φορτηγά. Γι' αυτό έχουμε μια πρώτη αναθεώρηση σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, τέσσερα χρόνια, γιατί θα έχουμε ήδη αρκετά στοιχεία. Το σπέκτρο με την ε, προσωμείωση που προσφέρει. Βέκτο. Το βέκτο με την ε, προσωμείωση που προσφέρει είναι ένα εργαλείο πρόοδου καθώς επιτρέπει στο μοντέλο αυτό να ενσωματώνεται κάθε νέα τεχνολογία όπως αυτή θα εμφανίζεται συν το χρόνο και έτσι μπορεί η Επιτροπή και θα έχει και πολλή δουλειά να επικαιροποιεί το βέκτρο για να καταγράφει τις νεότερες και πιο αποτελεσματικές τεχνολογίες. Έτσι και σε μία από τις προτινόμενες τροπολογίες που αναφέρεται στα πολύ μακριά φορτηγά, τα European Modular System Combinations, νομίζω ότι δεν θα έχουμε δυσκολία να τη δεχθούμε την τροπολογία αυτή. Υπάρχει όμως μια άλλη, η οποία έχει να κάνει με την ε, ε, απόσταση από την πηγή των καυσίμων στον τροχό, ε, πρέπει να κοιτάξουμε τι αποτελέσματα θα μας δώσει το σύστημα προσωμείωσης του βέκτου σε σχέση με τον ε, τομέα των καυσίμων, ο οποίος βεβαίως δεν είναι αρμοδιότητα της αυτοκινητοβιομηχανίας, ενώ η υποχρέωση την οποία βλέπουμε να καταγραφεί η τροπολογία επιβαρύνει την αυτοκινητοβιομηχανία. Πώς μπορεί λοιπόν η αυτοκινητοβιομηχανία να καταστεί υπεύθυνη για εκπομπές οι οποίες έχουν ε, ε, μπει στο σύστημα ήδη πριν το καύσιμο να μπει στην ε, δεξαμενή καύσιμο του αυτοκινήτου. Υπάρχουν και άλλα νομοθετήματα που θα πρέπει να σημειωθούν εδώ, όπως η οδηγία για τα νεώσιμα. Όταν ε, σχεδιάσαμε την ε, μείωση κατά, 30, κατά 40% των εκπομπών, το στόχο αυτό για την Ευρωπαϊκή Ένωση, είχαμε δεχθεί ότι θα πρέπει να συμβάλλουν και τα βαρέα φορτηγά. Ωστόσο, εάν υπολογίσουμε για δεύτερη φορά τα καύσιμα, με τα δύο καύσιμα μαζί, τότε επιβαρύνουμε το σύστημα χωρίς καμιά δυνατότητα να προχωρήσουμε. Και έτσι θα φτάσουμε το 2030 σε μείωση εκπομπών ε, στους 29 με 30 τόνους διοξιδίου του άνθρακα, χάρη στην ε, νομοθεσία των ανανεώσιμων, αλλά με το καινούριο αυτό νομοθέτημα και τη ρύθμιση των εκπομπών ε, για τα φορτηγά θα έχουμε μικρότερη μείωση. Έτσι λοιπόν, Εάν περιορίσουμε το πεδίο της νομοθεσίας θα ε, υποχρεωθούν οι, ε, θα υποχρεωθεί η αυτοκινητοβιομηχανία σε ουσιαστικά μηδενικές ε, αλλαγές ή μειώσεις των εκπομπών. Άρα πρέπει να υπολογιστούν και τα βιοκάψιμα. Είναι κάτι το οποίο θεωρούμε πάρα πολύ σημαντικό. Να μην υπολογίζονται οι εκπομπές των καυσαερίων ε, διαφορετικών νομοθετημάτων δύο φορές. Θα ήταν κακό, θα ήταν εσφαλμένο, θα σήμαινε επικάλυψη και επιβάρυνση γραφειοκρατική για την αυτοκινητοβιομηχανία, η οποία θα καλείτο να ε, κοινοποιεί, να ανακοινώνει τις εκπομπές αυτές, οι οποίες είναι εκτός των ε, δυνατοτήτων ελέγχου της και που ε, υπάρχουν στο σύστημα, ενσωματώνουν το σύστημα πριν να φτάσουν τα καύσιμα στο όχημα. Στο συγγνώμη που επιμένω σε αυτό, αλλά έχει μεγάλη σημασία και αυτό ανεξαρτήτως του αν είναι βαρέα τα οχήματα ή ελαφρά. Ευχαριστώ πολύ. Αυτό που είπατε με το Λουξεμβούργο λίγο με μπέρδεψε. Δευτέρα ψηφοφορία. Μυστική ψηφοφορία, τι είναι αυτό. Έτσι λοιπόν προχωρώ, δίνοντας το λόγο στο Δήμο, οπωσδήποτε για τα συμπεράσματα. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, ευχαριστώ τους σκιώδες εισηγητές για τόσα είπαν και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή βέβαια για την ξεκάθαρη παρουσίαση του ζητήματος αλλά απογοητεύτηκα κάπως από τους πράσινους, τον κύριο Νταλούντε, που λέει ότι δεν υπάρχει φιλοδοξία. Στο ΕΛΚ θεωρούμε ότι είναι μια πάρα πολύ φιλόδοξη πρόταση. Με τον Ταλούντεν το 2030 θα κοιτάξουμε να δούμε αν έχει πάει καλά ή όχι αυτή η υπόθεση. Ευχαριστώ. Καλώς, λέει ο πρόεδρος. Υπενθυμίζω ότι η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών είναι 13η Σεπτεμβρίου. Εμείς θα ψηφίσουμε στην Επιτροπή μας στις 9 Οκτωβρίου και περνάμε στο τελευταίο σημείο για σήμερα που είναι ο κανονισμός που προβλέπει πρώτος κανονισμού δηλαδή για τη θέσπιση διαστημικού προγράμματος της Ένωσης. Είναι γνωμοδότηση που ετοιμάζει η Επιτροπή μας για την Ήτρε. Οπότε, ο Βίμ στη θέση του κύριου Σαλίμη, που είναι η συγητής για αυτό το θέμα, το ΕΛΚ. Βίμ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Είναι σαφές, πέμπτη απόγευμα, όταν συνεδριάζουμε, ε, δεν έχουμε και πάρα πολύ επιτυχία. Σίγουρα, όταν υπάρχουν συνάδελφοι οι οποίοι έρχονται από μακριά και πρέπει να επιστρέψουν πίσω. Τέλος πάντων, αυτό το θέμα είναι ένα σημαντικό και πράγματι τη γνωμοδότηση του κύριου Σελήνη θα σας εξηγήσω. Διάστημα και μεταφορές έχουν άμεση σχέση σε, αυτό, σε αυτή την εποχή της τεχνολογίας που ζούμε. Τα διάφορα συστήματα μεταφορών συνδέονται μεταξύ τους αλλά και η διαχείριση των μεταφορών είναι πράγματα που συνδέονται με τις διαστημικές υπηρεσίες. Και το ERTMS, που είναι το δίκτυο ασφάλειας στη θάλασσα, επίσης συνδέεται με τις διαστημικές αυτές υπηρεσίες. Και υπάρχει βέβαια και η οικονομία του διαστήματος. Βέβαια, θέλω να πω ότι υπάρχουν και τα αυτόνομα οχήματα, αλλά υπάρχει και το κλίμα και η κλιματική αλλαγή που μπορεί να επωφεληθεί από μια καλή διαστημική βιομηχανία στην Ευρώπη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν έχει τον Κοπέρνικο, το Γαλιλαίο και το Έγνος και τα τρία μαζί θα τεθούν σε εφαρμογή που είναι προγράμματα δορυφορικής πλοήγησης και θα αποτελέσουν ένα πρόγραμμα. Αυτό που είναι σημαντικό πρόεδρε εδώ στα πλαίσια του νέου πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου να υπάρχουν αρκετά χρήματα για την περίοδο 2021 με 2027. Και είναι πολύ σημαντικό ο διαστημικός τομέας να βοηθήσει και να εξυπηρετήσει ώστε και οι οδικές μεταφορές και θελάσσιες και αεροπορικές να γίνουν περισσότερο ασφαλείς και περισσότερο βιώσιμες. Η υπηρεσία λοιπόν για τα διαστημικά προγράμματα όλα αυτά θα πρέπει να τα έχει υπόψη της, να τετικοποιήσει τις προσπάθειές της και να μπορέσει να βοηθήσει όλες τις μορφές μεταφορών. Ο κύριος Σαλίνη λοιπόν επιμένει στη διαστημική μας υπηρεσία και υπογραμμίζει και το θέμα των ε, δορυφόρων που δεν χρησιμοποιούνται πια, που έχουν καταστραφεί. Και συμφωνώ και εγώ ότι πρέπει να δούμε τι γίνεται με όλους αυτούς οι οποίοι κυκλοφορούν στο διάστημα. Μην αρχίσει και βρέχει παλιούς δορυφόρους ή κομμάτια τους. Υπάρχει και το πρόγραμμα satellite.com και εδώ πρέπει να ξέρουμε αυτή η διευκόλυνση τι ρόλο ακριβώς θα παίξει στις μεταφορές. Τέλος, Πρόεδρε, το θέμα της κυβερνοασφάλειας γιατί όλες αυτές οι τεχνολογικές εξελίξεις μπορεί να τύχουν κατάχρηση από κακόβουλους. Πρέπει συνεπώς να υπάρχει προστασία τους. Ο κύριος Αλήνη λοιπόν λέει ότι το πρόγραμμα αυτό είναι ανεξάρτητο βέβαια, αλλά υπάρχει ανταγωνισμός και πρέπει να μπορούμε να συνεργαζόμαστε με τους εταίρους μας και μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εκτός. Πρόεδρος, ευχαριστούμε Δήμ. Και το λόγο θα πάρει κύριε Νταλόν, η οποία είναι σε One Woman Show απόψε. Α, όχι, όχι εσύ. Ω, συγγνώμη, μπέρδεψα τις κυρίες. Θα στήσει το λόγο μας μετά. Μάλιστα, καλώς. Κύριε το λοιπόν, και Εκ μέρους του κύριου Ασής, Πρόεδρε. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω τον ε, εισηγητή για τα όσα μας είπε. Έχουμε να κάνουμε ένα πολύ σημαντικό για το χώρο των μεταφορών ε, ζήτημα. Η επιστημονική έρευνα των πόρων αυτών μας δείχνει ότι υπάρχει μια σειρά από ευκαιρίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κράτη-μέλη, τη βιομηχανία, τους πολίτες και είναι οι προκλήσεις που αντιμετωπίσουμε, η κλιματική αλλαγή, η βιώσιμη ανάπτυξη, η αυτόνομη οδήγηση, οι, οι γνωστές ήδη, η ασφάλεια, η άμυνα, λίγη των συνόρων, ε, ασφάλεια οδική. Είναι προκλήσεις που μπορούν να βρουν ένα νέο πεδίο ε, και πρέπει να είμαστε στην πρώτη καθεδρία στη διερεύνηση αυτού του πεδίου. Και βεβαίως χαίρομαι που καθίσατε μια από τι προτεραιότητε τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η διερεύνηση του διαστήματο. Χρειαζόμαστε περισσότερους πόρου για την έρευνα και την ανάπτυξη. Το ΕΠΕΦ, πολιτιστικό νομικό πλαίσιο που έχει προτείνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, κατά την απόψή μα δεν είναι αρκετά φιλόδοξο. Πρέπει να επιδιώξουμε περισσότερου ευρωπαϊκού πόρου προκειμένου να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα που έχουμε στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Και θα ήθελα κλείνοντα να πω ότι η ομάδα μου θα συμβάλλει στην συζήτηση με ορισμένε τροπολογίε και ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να συνεργαστούμε και να καταλήξουμε σε ένα πολύ καλό κείμενο εν τέλει. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Ντεόντε. Και θα εκπροσωπήσω τον κύριο Τζέλισκα, τον οποίο κάλεσε ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου σε μια άλλη εκδήλωση, σκιώδης ηγητή της ομάδας μου. Ο Στελίτσκα θα ήθελα να ευχαριστήσει τον εισηγητή για την προτάση σας προς τον κανονισμό με τις οποίες συμφωνεί σε μεγάλο βαθμό. Σε ό,τι αφορά το σχετικά ε, σύντομο χρονοδιάγραμμα για το πιδελταπή, συμφωνεί με τον εισηγητή σε ό,τι αφορά την συμπίκνωση των εργασιών μας και την επικέντρωση σε μικρό αριθμό στρατηγικών προτεραιοτήτων σε ό,τι αφορά το γενικό προϋπολογισμό. Είναι υπερ ε, ε, του προγράμματος για τις διάφορες δραστηριότητε στο, στο διαστημα, στον τομέα του διαστήματος, προκειμένου να έχουμε μια συνεκτική ευρωπαϊκή στρατηγική. Ε, κάτι που θα διευκολύνει την παρακολούθηση και την εφαρμογή της κατά την περίοδο 2021-2017 και οι συνέργειες που ενθαρρύνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με το ενιαίο διαστημικό πρόγραμμα δεν θα παραμείνουν στο επίπεδο αγαθών προθέσεων μόνο. Επίσης, ο κύριος Τελίσκα είναι σαφώς υπέρ ε, διεύρυνσης της εντολής ε, του οργανισμού που έχει έδρα ε, στην Πράγα. Είναι σημαντικό το έργο του προγράμματος αυτού και για τις μεταφορές και είναι σημαντικό η Επιτροπή ΤΡΑ να αποφανθεί με νέα φωνή και να δοθεί σάρκα και ωστά στο πρόγραμμα αυτό κατά την επόμενη περίοδο προγραμματισμού. Και με αυτή την άποψη ο κύριος Τελίτσκα θα επικεντρωθεί σε τέσσερις κυρίως προτεραιότητες. Πρώτον, εξασφάλιση επαρκούς προϋπολογισμού με βάση τη σημασία που έχει το πρόγραμμα ε, για τον τομέα των μεταφορών ε, και επίσης οι πόροι που προβλέπονται θα πρέπει να καλυφθούν και δημοσιονομικά σε ό,τι αφορά την κατανομή των κονδυλίων μεταξύ των προγραμμάτων και των οργανισμών, αλλά και σε αλληλεπίδραση με άλλα προγράμματα. Επίση θα πρέπει να σε τεχνο... να εξασφαλιστεί η πρόσβαση στις τεχνολογίες που θα ε, αναπτυχθούν με βάση το πρόγραμμα και επίσης ε, να καταλήξουμε σε πρότυμα και προδιαγραφές, ε, προδιαγραφές με βάση αυτές τις νέες τεχνολογίες. Επίσης, τονίζουμε την κυβερνοδιάσταση που έχει ένα τέτοιο διαστημικό πρόγραμμα. Και μάλιστα ε, θα πρέπει να συνεχίσουμε τη συζήτηση για την εντολή της ΕΝΗΣΑ. Επίσης, θα πρέπει να εξασφαλίσουμε αξιολόγηση του προγράμματος και των αποτελεσμάτων. άλλωστε, όλα αυτά τα είχε πει ήδη ο κύριος Τελίτσκα στα πλαίσια της συζήτησης ε, για την ε, ε, σύνδεση, την ε, σύνδεση στην Ευρώπη, το σύστημα MIE, το Μηχανισμό Διασύνδεσης Ευρώπης. κυρία Ρεβόνταλόν, ευχαριστώ. Χαιρετίζω το αξιόλογο έργο του εισηγητού που είναι και σε πολιτικό και σε ουσιαστικό επίπεδο πολύ χρήσιμο για την επόμενη περίοδο προγραμματισμού και το διαστημικό πρόγραμμα. Και μάλιστα ε, ευθυγραμμίζεται με τις προτεραιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπως φαινόταν στις προτεραιότητες για την διαστημική στρατηγική, προκειμένου να ε, εφαρμοστεί στον τομέα των μεταφορών ε, εφαρμογές αυτού του προγράμματος Και ελπίζω να ληφθούν υπόψη οι προτάσει του εισηγητού μια ναι, και ο κύριο Σελήνη είναι ο εισηγητή για το ίδιο θέμα και στην Ήτρε, κάτι που θα διευκολύνει πολύ τη συνεργασία μεταξύ των δύο επιτροπών. Συμφωνώ με τι τροπολογίε που είναι υπέρ τη ευρωπαϊκή προτίμηση για τι θεσμικέ ε, ε, αγορές ό,τι αφορά τους εκτοξευτήρες δορυφόρων. Επίσης, αυτό είναι ένα πολύ ιδιαίτερο πρόβλημα που θα πρέπει να ληφθεί υπόψη στη διαστημική μας στρατηγική και μάλιστα θα καταθέσω τροπολογίες για να εμπεδώσουμε αυτή την ευρωπαϊκή προτίμηση σε ένα στρατηγικό τομέα που έχει σχέση με την κυριαρχία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί περί αυτού πρόκειται να μιλούμε για πρόσβαση στο διάστημα. Ο κανονισμός προβλέπει την ε, θέσπιση προγράμματος εργασίας για την επόμενη 20 ετία για την εκτόξευση δορυφόρων. Γιατί αυτό ήταν το αίτημα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και θα ήθελα να μου πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε τι φάση βρίσκεται σε αυτόν τον κανονισμό. Ευχαριστούμε. Έχω να κάνω και κάποιες προσωπικές παρατηρήσεις. Η ποιότητα του προτινόμενου κανονισμού είναι ε, αντίστοιχη της ποιότητα του κειμένου του εισηγητή. Είναι ένα θέμα που έχει να κάνει με την ευρωπαϊκή κυριαρχία, έτσι, πολύ σημαντικό. Δεν υπάρχει διαστημική πολιτική στη σωστή κλίμακα, υπάρχει σε επίπεδο χωρών μελών. Αλλά αν δεν υπάρχει σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα είμαστε τρίτης κατηγορίας. Και μπορούμε να αναρωτηθούμε τι θα γινόταν με την κυριαρχία της Ευρώπης αλλά ακόμα και των χωρών μελών και κάποιων που θέλουν αυτόνομη άμυνα αν δεν γινόταν αυτή η ευρωπαϊκή προσπάθεια. Οπότε μπορεί να υπάρχει θέμα κυριαρχίας για τις χώρες μέλη, αλλά ακριβώ αυτό συζητάει η έκθεση. Και κάποιες άλλες παρατηρήσεις. Το θέμα αυτό σέβεται ε, το ζήτημα των εκτοξευτών, που είναι ένα πολύ ευαίσθητο θέμα για να ξαναρχίσει το πρόγραμμα Ριάν 6 και βλέπουμε τις στρατηγικές δυσκολίες δεδομένες της εξέλιξης της πολιτικής εκτοξευτών, κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου περνάει στα χέρια του ιδιωτικού τομέα. Πρέπει οπωσδήποτε να μείνουμε και εμείς σε αυτόν τον αγώνα, να είμαστε παρόντες και άρα πρέπει να ξαναδούμε το δημοσιονομικό ζήτημα της χρηματοδότησης δηλαδή, για να έχουμε αρκετά χρήματα, γιατί αλλιώς θα χάσουμε πλήρως τον αγώνα αυτών. Δεύτερον, σε αυτά τα πλαίσια είναι πολύ σημαντικό να έχουμε ένα πολιετές πρόγραμμα αφιερωμένο στους ευρωπαϊκούς εκτοξευτές. Είναι πολύ σημαντικό δεδομένη της δέσμευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και υπάρχει και το downstream, δηλαδή υπάρχουν πολύ περισσότερα χρήματα για την εκμετάλλευση δεδομένων που μας έρχονται από το διάστημα από ότι ε, στους μηχανισμούς που χρειαζόμαστε για να αποκτήσουμε αυτά τα δεδομένα. Οπότε πρέπει να μας απασχολήσει αυτό και να ευνοήσουμε τις επιχειρήσεις εκείνες οι οποίες μας βοηθούν να κερδίσουμε περισσότερα από τις διαστημικές υπηρεσίες. Αυτές είναι οι παρατηρήσεις μου. Φυσικά και θα στηρίξουμε. Και εγώ προσωπικά θα υποβάλω κάποιες τροπολογίες. Πάντως αυτό το θέμα είναι πολύ σημαντικό. Τώρα, η κυρία Κονέσκα από την ΚΟΕ. Παρακαλώ. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρε, ήθελα και εγώ να πω δύο λόγια για το έγγραφο αυτό. Θα ήθελα να πω ότι αντίθετα από σας η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με απογοήτευσε. Λυσμονήθηκε τελείως η ανάγκη να γίνει πιο φθηνή, πιο γρήγορη η υλοποίηση της, του προγράμματος. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν θα έχει να διαχειριστεί ένα πρόγραμμα ε, χωρίς όμως να λαμβάνει υπόψη τις ε, αρμοδιότητες που ε, πρέπει να είναι να ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος. Δεν μπορεί να ελέγξει τις δραστηριότητες αυτές και πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να διαδραματίσει το ρόλο μιας αρχής επιδιαιτησίας σε σχέση με τη χρήση των κονδυλίων, σε σχέση με τη ρύθμιση της δραστηριότητες και τα τεχνικά ζητήματα. Η ΕΣΑ λοιπόν θα είναι, ε, θα στηρίζεται στην, επιτεχνο, στην επιδιατησία της Επιτροπής η οποία ε, ΕΣΑ θα περιορίζεται μόνο σε τεχνικά ζητήματα. Η πρόταση δεν δίνει αποτελεσματικές λύσεις και με τις τροπολογίες μας θα προσπαθήσουμε να αντιμετωπίσουμε τις δυσκολίες. Ευχαριστώ. Euh, για την πολιτική για το διάστημα είναι απαραίτητο αυτό οπωσδήποτε και δίνω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κύριε Ντέλσο, έχετε το λόγο. Να, το βρήκα, το βρήκα. Δουλεύει. Ε, το πρόγραμμα για το διάστημα δουλεύει καλύτερα από τα μικρόφωνά σας. Δεν είναι και δύσκολο. Ένα θα συμπληρώσω μόνο στα όσα είπα πριν, αυτό που υπογραμμίσατε και εσείς Πρόεδρε, ότι δεν θα ήταν δυνατό αυτό που κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση να το κάνουμε μόνο με ένα τα κράτη-μέλη. Αν κοιτάξουμε το πρόγραμμα Γαλιλαίους, οπωσδήποτε ενδιαφέρει πολύ την Επιτροπή σας, μας επιτρέπει ήδη αυτή τη στιγμή που μιλάμε ακρίβεια που κανένα άλλο πρόγραμμα του κόσμου δεν εξασφαλίζει. Το Γαλιλαίος δηλαδή ήδη θεωρείται πως είναι πολύ πιο επιτυχημένο από οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα γεωεντοπισμού. Νομίζω ότι οφείλουμε μερικές φορές να αναγνωρίζουμε και να είμαστε υπερήφανοι για αυτά τα οποία κάνουμε από κοινού. Το ίδιο και για το Κοπέρνικος, το οποίο πολλοί θεωρούν πως έχει επιτύχει εξαιρετικά αποτελέσματα με ένα παράδειγμα που θα σας δώσω. Το Υπουργείο Εξωτερικών μεγάλης χώρας ε, πέραν του Ατλαντικού, εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που συχνά ε, υποβλέπει τις λοιπές χώρες και υπηρεσίες του, ε, ζήτησε από το Κομπέρνικο υπηρεσίες, από το Γαλιλαίος υπηρεσίες για να μπορέσει να αντιμετωπίσει μεγάλη φυσική καταστροφή που είχε εγκύψει. Ε, θα ήθελα λοιπόν τώρα να ευχαριστήσω τον εισηγητή και την Επιτροπή σας για όλη τη δουλειά. Μια σειρά από παρατηρήσεις είναι πολύ σημαντικές. Η πολιτική, η σχετική με τους εκτοξευτές είναι πάρα πολύ σημαντική. Εδώ το ζήτημα της ευρωπαϊκής αυτονομίας και είναι πολύ σημαντικό στο κείμενο το οποίο έχουμε προτείνει να αποστελέτε ένα σαφές μήνυμα για την πολιτική αυτή. Οπωσδήποτε ε, αναγνωρίζουμε ότι είναι διφιλονικούμενο το ζήτημα, αλλά είναι σημαντικό να διατυπώσουμε προτάσεις και το Κοινοβούλιο επίσης. Έχουμε καταθέσει προτάσεις μας και ελπίζουμε ότι θα μπορέσει να ε, τύχει της υποστήριξης του Κοινοβουλίου στο σύνολό του. Ε, δυστυχώς για την μακροπρόθεσμη πολιτική και το στρατηγικό όραμα των προσεχών 20 ετών, Δυστυχώ, οι περιορισμοί που αντιμετωπίζουμε είναι αυτοί των πιο σύντομων δημοσιονομικών κύκλων, που μας ε, δεσμεύουν. Δηλαδή το πολιτισμικό πλαίσιο ε, είναι αυτό που είναι, είναι μόνο επταετές και ως εκ τούτου δεν μπορώ να αναλάβω δέσμευση άλλη από αυτή την οποία έχουμε ήδη μέσα στη στρατηγική για το διάστημα που έχει άλλωστε εγκρίνει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ε, διακυβέρνηση, πολύ λεπτό πάντα θέμα, αλλά θα ήθελα να σας καθησυχάσω. Η Επιτροπή δεν σκοπεύει να πεμπολίσει τις ε, ευθύνε της. Είμαστε αποφασισμένοι, θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με βάση ευθύνε που έχουμε αναλάβει. Σε τελευταία ανάλυση ε, είναι σημαντικό να έχουμε συμφωνία μεταξύ όλων των παραγόντων της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Διαστήματος, της δικής μας υπηρεσίας, το διάστημα και βέβαια τη Επιτροπή για μια ε, καλή και αρμονική συνεργασία. Το χειρότερο που θα μπορούσε να συμβεί ήταν να διχαστούμε εμεί οι Ευρωπαίοι μεταξύ μα. Αν δεν μπορέσουμε να συνεργαστούμε δηλαδή κατά τρόπο εναρμονισμένο μεταξύ μα, κινδυνεύουμε να μην μπορέσουμε να διαφυλάξουμε την πρωτοκαθεδρία αυτή που έχουμε σε επίπεδο τόσο Γαλιλαίου όσο και Κοπέρνικου. Τέλο, και γενικά ω θεώρηση για το μέλλον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν σκοπεύει να κάνει καμία επανάσταση. Θέλει να βελτιώσει αυτά που υπάρχουν. Θέλει να εξασφαλίσει ότι τελικά θα, μπορούσε, θα μπορούμε να έχουμε κάποια προγράμματα που σε 10 χρόνια ο διάδοχό μου που θα έρθει να σα μιλήσει εδώ στο Κοινοβούλιο θα είναι πάλι σε θέση να σα καθησυχάσει, να σα διαβεβαιώσει ότι το πρόγραμμά μα είναι το καλύτερο στον κόσμο. Ή τα προγράμματά μα είναι τα καλύτερα στον κόσμο. Αυτά. Και τα είπε πολύ ωραία, λέει ο Πρόεδρο. Βήμα. Ξέρω, θα σου το λόγο, αλλά πριν νομίζω ότι μια και ο κύριος Τέιλορ ήρθε εγκαίρος, του δίνω το λόγο και τι δεν ήθιστε να λαμβάνουμε το λόγο όταν έχει μιλήσει ο εκπρόσωπος της Επιτροπής, αλλά μια και έχουμε και ένα μεγάλο χρονικό περιθώριο, έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ. Δεν μπορώ να υποκρίνομαι ότι είναι ε, ειδικότητά μου αυτό αν εξαρτάται από μένα θα διάλεγα άλλο θέμα. Δεν είχα και μεγάλη εξοικείωση με τα θέματα του διαστήματος. Πάντως θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Σαλίνη για το έργο του σε ό,τι αφορά αυτό το διαστημικό πρόγραμμα. Και ουσιαστικά ενισχύω με αυτά που είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ότι το διάστημα είναι η κοινή μας κληρονομιά που θα πρέπει να τη διαφυλάξουμε και για τις επερχόμενες γενές και θα πρέπει να ενθαρρύνουμε υπεύθυνη συμπεριφορά στο διάστημα και εκτός του, πέραν του διαστήματος. Εκ μέρους των Πρασίνων θα υποβάλουμε κάποιες τροπολογίες για την βιωσιμότητα προκειμένου να αποτρέψουμε μία κούρσα που θα εξαντλήσει τους σπόρους μας. Επίσης θα συμπεριλάβουμε και την ανάγκη αποτελεσμάτων των υπηρεσιών Γκαλιλαίο και Κοπέρνικος που θα πρέπει να προσφέρονται δωρεάν σε άλλες ενδιαφερόμενες αρχές και θα ζητήσουμε αύξηση της στήριξη για τα καινοτόμα συστήματα και την ανάπτυξη καινοτόμων υπηρεσιών. Επίσης, θα θέλαμε βελτίωση και στα θέματα ισότητας των φύλων στον τομέα του διαστήματος, εξασφαλίζοντας ε, η συμμετοχή στα διοικητικά συμβούλια να τηρούν την ισορροπία μεταξύ των δύο φύλων. Προσβλέπω σε αγαστή συνεργασία με τον εισηγητή και τους κοιόδης εισηγητές ε, τις επόμενες εβδομάδες και μήνες. Σας ευχαριστώ που μου δώσετε την ευκαιρία, κύριε Πρόεδρε, να λάβω το λόγο. Ε, ε, ευχαριστώ. Και ο τελευταίος λόγος των Βίμ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Είναι βέβαια φοβερό από ολόκληρη αυτή τη μεγάλη ομάδα που είναι το ΕΛΚ να έχω αναλάβει εγώ τέσσερις εκθέσεις. Πάντως ευχαριστώ πολύ τους και όδους και πάλι για τα όσα είπαν. Ευχαριστώ πολύ και για την ξεκάθαρη παρουσίασή της στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα ενημερώσω τον κύριο Σαλίνη. Σίγουρα μέσω διαδικτύου θα έχει παρακολουθήσει ο κύριο Σαλβίνη και θα έχει σημειώσει όλες ε, τις παρατηρήσεις και τα σχόλιά σας. Και στον κύριο Τέιλορ θέλω να πω ευχαριστώ πολύ. Έχουμε εδώ και γυναίκες. Είμαι σίγουρος ότι υπάρχει μεγάλη ποιότητα σε όλα τα σχόλια που ακούσαμε. Ευχαριστώ πολύ. Με αυτά τα λόγια, λέει ο Πρόεδρος, γεμάτα κοινή λογική, ολοκληρώνουμε τη συνεδρίασή μας για σήμερα. Η επόμενη... Α, όχι, μια στιγμή. Προθεσμία για υποβολή τροπολογιών 5η 13 Σεπτεμβρίου στις 12 το μεσημέρι. Δηλαδή πριν πάτε να φάτε εκείνη την ημέρα, μην ξεχάσετε να υποβάλλετε τις τροπολογίες σας. Επόμενη συνεδρίαση 24 Σεπτεμβρίου 2018. Ολοκληρώσαμε για σήμερα, λίγο νωρίτερα από το προκαθαρισμένο και επειδή οι παρόντες συνεργάστηκαν τόσο καλά, αλλά και επειδή οι απόντες ήταν τόσο πολύ. Αυτά. Καλό βράδυ σε όλους. Ξεχάστε τον αγώνα ποδοσφαίρου 20 και 45. Κλασικό.